So, ladies and gentlemen, it's minutes past I would like... Λοιπόν, έχει ε, περάσει η ώρα. Είναι σχεδόν 10 και 10. Θα ήθελα να αρχίσουμε. Συνεδρία τη Επιτροπή Εξωτερικών. Ζητώ συγγνώμη για τη χθεσινή μου απουσία. Αλλά έπρεπε να εκφωνήσω ένα λόγο. Στην κάτω Σαξονία για ένα ε, πρώην υπουργό αλλά έμαθα ότι προέδρευσε ο κύριο Βίστησεν και πήγαν όλα καλά. Ε, σημείο 14. Θα ήθελα να καλωσώσω τον Ζίκφριτ Μούρεσαν, αγαπητέ Ζίκφριτ, καλώς όρισε, εισηγητή τη Επιτροπή Προπολογισμών για τον Προπολογισμό 2018 τη Ευρωπαϊκή Ένωση, για να συζητήσουμε τι προτεραιότητε για τι δαπάνε Ευρωπαϊκή Ένωση του 2018. Όπω κάθε χρόνο η Επιτροπή μα ε, γνωμοδοτεί και ψηφίζει ε, τι τροπολογίε τη τον Αύγουστο θα επικεντρωθούμε στις δαπάνες για την εξωτερική δράση του τίτλου 4 του πολιετούς ε, δημοσιονομικού πλαισίου. Θα πρότεινα να δώσω το λόγο τώρα στο Ζικβιτμού και μετά στο συντάκτη γνωμοδότησης της δικής μας επιτροπής, τον Κρίστιαν Πρέντα. Έχεις το λόγο, Ζικβιτ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που με υποδέχεστε όλοι εδώ. Ευχαριστώ τους συναδέλφους θα ήθελα να μου επιτρέψετε να σας παρουσιάσω τις βασικές πολιτικές προτεραιότητες του προϋπολογισμού της Ένωσης, οι οποίες υιοθετήθησαν από την Ολομέλεια με μεγάλη πλειοψηφία τον μήνα Μάρτιο. Δεύτερον, και αυτό ίσως είναι πιο σημαντικό, ήρθα να ακούσω από εσά τις συγκεκριμένες προτεραιότητες, τα επιμέρους προγράμματα, τα οποία θα πρέπει να πληκίσουμε με τον επαρκή προϋπολογισμό για τα επόμενα χρόνια. Θα ήθελα λοιπόν η παρουσία μου εδώ σήμερα να είναι η αρχή μιας μακράς συνεργασίας. Όπως είπα, οι κατευθυντήριες γραμμές έχουν γίνει δεκτές για τον επόμενο χρόνο. Περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει την πρόταση προϋπολογισμού στο τέλος Μαΐου και στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων που θα κάνουμε με την Επιτροπή και το Συμβούλιο έχει σημασία για μένα να γνωρίζω την δική σας άποψη για την πρόταση την οποία κάνει η Επιτροπή και πιθανώς να διευκρινίσετε κι εσείς από πλευρά σας τις ε, τροπολογίες ε, οι οποίες σας ενδιαφέρουν και να ακούσω επίσης και τις προτάσεις του κυρίου Πρέντα. Τώρα για τις βασικές πολιτικές προτεραιότητες. Υπάρχουν δύο βασικές τέτοιες προτεραιότητες. Πρώτον, ανάπτυξη θέσης απασχόλησης και δεύτερον, ασφάλεια των πολιτών. Νομίζω ότι αυτό περιμένουν από εμά οι πολίτες, να χρησιμοποιούμε τον προϋπολογισμό για θέσεις εργασίας και δεύτερον για ασφάλεια. Πώς μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Πρώτον θα πρέπει να υποστηρίξουμε τη διαδικασία δημιουργίας θέσεων εργασίας μέσω μιας καλύτερης οικονομίας, μιας πιο ισχυρής οικονομίας, ελκυστικής για τον ιδιωτικό τομέα και τους επενδυτές. Λοιπόν, υποδομές, έρευνα και ανάπτυξη, υποστήριξη των μικρομεσαίων, υποστήριξη των νέων επιχειρηματιών, και στα πλαίσια του Horizon 2020, του Connecting Europe, του COSME και το Erasmus που δεν είναι ένα πρόγραμμα μόνο για φοιτητέ, αλλά όπως ξέρετε το 60% των εργοδοτών όταν προσλαμβάνουν κάποιον ε, θεωρούν θετικό πράγμα την ε, ε, διαδικασία Erasmus. Πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε σωστά τα μέσα αυτά για να βρουν οι νέοι σωστές θέσεις εργασίας καλά αμοιβόμενε. Τώρα για την ασφάλεια των πολιτών, που έχει σημασία νομίζω ιδιαίτερη για σας. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πετύχουμε πρώτον, όπως γνωρίζετε, οι πόροι που έχουμε στο 3 και στο 4 είναι περιορισμένοι. Πώς μπορούμε λοιπόν να πετύχουμε περισσότερα με τους ε, ελαχιστοποιημένους πόρους. Και δεύτερον, Είμαι υπέρ της προπαρασκευαστικής δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα της άμυνας. Πέρυσι ήμουνα σκιώδης εξ ονόματος της πολιτικής μου ομάδας για τον προϋπολογισμό για το 2017. Υποστήριξα την προπαρασκευαστική δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις κατευθυντήριες γραμμές τώρα στις οποίες, τις οποίες υιοθετήσαμε στην Ολομέλεια. Στηρίζουμε κάθε πρωτοβουλία στον τομέα της έρευνας και της άμυνας γιατί απαιτείται να υπάρχει συνέχεια, να αποφύγουμε επικαλύψεις, να μην ξοδεύουμε 28 φορές τα ίδια χρήματα για, τα ίδια, για τους ίδιους στόχους και να συνεργαζόμαστε και στα πλαίσια άλλων σχημάτων όπως το ΝΑΤΟ. Η έκθεσή μου λοιπόν είναι σαφής, ζητώντας μια ξεχωριστή δημοσιονομική γραμμή για το επόμενο πολιετές ε, στα πλαίσια της άμυνας και της έρευνας για την άμυνα. Οι προτάσεις μέχρι τώρα δεν είναι κακές, αλλά είναι μια απλή αρχή και πρέπει να ενισχυθούν. Για να πετύχουμε μεγαλύτερη ασφάλεια λοιπόν έχουμε πρώτον την προπαρασκευαστική δράση, δεύτερον να ενισχύσουμε τις εξωτερικές υπηρεσίες που είναι υπεύθυνε όπως η Frontex, η Eurojust, η ASO, Αυτά οδηγούν στην καλύτερη προστασία των συνόρων μας, στην καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών για την καταπολέμηση φαινομένων όπως το λαθρεμπόριο όπλων, η τρομοκρατία και το σωματεμπόριο. Μια ασφαλέστερη λοιπόν Ευρώπη. Αυτό είναι σημαντικό και για την ανατολική γειτονία. Βλέπουμε μια πιο δραστήρια ρωσική ομοσπονδία, μια πιο επιθετική αν θέλετε πρόεδρε, και αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν προκλήσεις εκεί και προκλήσεις υπάρχουν και στη νότια γειτονία. Πρέπει να στηρίξουμε λοιπόν τις χώρες στην ανατολική γειτονία που ακολουθούν την ευρωπαϊκή γραμμή έχοντας υπογράψει και επικυρώσει εταιρικέ συμφωνίες με την Ένωση. Γεωργία, Ουκρανία και Μολδαβία θα πρέπει να τύχουν μεγαλύτερης οικονομικής ενίσχυσης, στα πλαίσια βέβαια μια αυστηρής αιρεσιμότητας με βασικό στόχο την ενίσχυση των θεσμικών του οργάνων, την καταπολέμηση της διαφοράς, βελτίωση του κράτους δικαίου, της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, της έκπληξης βρώμικου χρήματος κτλ. Αυτά για την ανατολική γειτονία, ιδιαίτερα για τις χώρες στις οποίες αναφέρθηκα και μετά υπάρχει και η νότια γειτονία. Πέρυσι το Μάιο με την Επιτροπή Προϋπολογισμών επισκεφθήκαμε την Ιορδανία και το Λίβανο και είδαμε ότι μπορούμε να πετύχουμε πολύ περισσότερα υποστηρίζοντας τους πρόσφυγες στην περιοχή τους, παρότι στο εσωτερικό της Ένωσης και κοστίζει λιγότερο και είναι πολιτικά πιο εύκολο και ασφαλέστερο αυτοί οι οποίοι έχουν ανάγκες να παραμένουν κοντά στις αιστείες τους. Και δεν αρκεί το να λένε στο Λίβανο και στην Ιορδανία ότι όταν τελειώσει η σύραξη θα επιστρέψουν στη χώρα τους. Πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε. Σχετικά τώρα με τα καταπιστεύματα, Ξέρετε ότι όταν δημιουργήθηκαν, είπαμε στην Επιτροπή Προϋπολογισμών ότι τα χρειαζόμαστε, είναι χρήσιμα, αλλά δεν μας αρέσει καθόλου ότι μάθαμε από το Κοινοβούλιο ότι θα πρέπει να δώσουμε 500 εκατομμύρια από τον κοινοτικό προϋπολογισμό στο μέσο για την Τουρκία. Κάναμε αυτό που έπρεπε βέβαια, αλλά δώσαμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι ε, αυτή τη φορά λόγω του κατεπήγοντος χαρακτήρα της υπόθεσης ε, το δεχτήκαμε, αλλά θα πρέπει να εμπλακούμε και στην φάση προετοιμασίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν τώρα μας ενημερώνει τακτικά για το στάδιο της εφαρμογής, για την κατάσταση της εφαρμογής των συμφωνιών αυτών και θα προσκαλέσει και εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, στα διοικητικά συμβούλια αυτών των καταπιστευμάτων. Αλλά το πρόβλημα παραμένει. Για το ε, Ταμείο Μαντάτ, σαν παράδειγμα, εμείς είχαμε ε, προβλέψει 1,1 δις από τον προϋπολογισμό της Ένωσης ενώ τα κράτη-μέλη από τις δικές τους υποχρεώσεις ε, επέλεξαν να δώσουν μόνο 117.000. Μία τελευταία παρατήρηση για την αναθεώρηση του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Αν προχωρήσουμε νομίζω ότι θα κερδίσουμε όλοι γιατί όταν αποφασίστηκε το πολιετές το 2013 για την περίοδο 14-20 δεν είχαμε προβλέψει ούτε την κρίση των προσφύγων, ούτε τα προβλήματα ασφάλειας και τρομοκρατίας. Πρέπει να ε, αποδώσουμε καλύτερα, να κάνουμε περισσότερα. Εμείς ε, ωφελούμεθα από την αναθεώρηση του πολιετούς κατά 1,5 δις και 750 στα πλαίσια της εταιρικής διαδικασίας, για την ΚΕΠΑ επίσης και την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, 274 για το ELM, την Ευρωπαϊκή επίσης Τράπεζα Επενδύσεων και 200 κάτι για, την, για θέματα ενισχύσεων και τις λεγόμενες micro assistance. Εμείς λοιπόν κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνει, εγκρίναμε τις αποφάσεις τις οποίες έπρεπε να πάρουμε, καταλήξαμε γρήγορα. Το Συμβούλιο έπρεπε να υιοθετήσει την προηγούμενη εβδομάδα στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων το, τη νέα πρόταση για το δημοσιονομικό πλαίσιο, το πολιετές, αλλά λόγω των εκλογών στην Αγγλία θα καθυστερήσουμε. Λοιπόν, η καθυστέρηση για λίγους μήνες δεν είναι ένα πρόβλημα. Αν τα υιοθετήσουμε τον Ιούλιο, είναι αρκετός ο χρόνος που θα έχουμε μετά. Αν όμως δεν γίνει κάτι τέτοιο τον Ιούλιο, τότε ο προϋπολογισμός για τον επόμενο χρόνο θα είναι πολύ δύσκολος. Δεν θα μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε αυτά τα οποία προγραμματίζαμε, αλλά και σε άλλους τομείς. Σαν παράδειγμα, αύξηση του κόσμου για 120 εκατομμύρια, και μάλιστα εμείς ζητήσαμε 200 εκατομμύρια για το κόσμο και τις μικροπεσαίες. Πώς θα το πετύχουμε αυτό λοιπόν. Ε, και μάλιστα ε, το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να ωφεληθεί και αυτό γιατί θα παραμένει τότε μέλος ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι λογικό αυτό γιατί τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν ηγετική θέση παγκόσμια. Λοιπόν, ε, εσείς στείλατε τα, τις δικές σας προτεραιότητες ή μάλλον ήταν η προθεσμία μέχρι σήμερα στις 12 το μεσημέρι. Όλα αυτά θα τα στείλουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να τα επανεξετάσει και θα αποφασίσουμε εκ των υστέρων από κοινού για ένα πακέτο χρηματοδότησης το οποίο θα βασίζεται στις δικές σας προτάσεις ε, για τις οποίες όπως είπα θα περιμένουμε το σχόλιο της Κομισιόν. Σας ευχαριστώ για μια ακόμη φορά που με δεχτήκατε εδώ και περιμένω τις απόψεις σας ε, και την γνωμοδότηση του κυρίου Πρέντα. Thank you, Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε τον Siegfried Μουρισάν για τα σχόλια αυτά και τώρα θα ακούσουμε τον σκιώτη συγκεκριτή μας ή τον εισηγητή. Συγγνώμη, συγγνώμη. Από πλευρά τη Επιτροπή ε, ΑΦΕΤ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Και καταρχά θα ήθελα να καλωσορίσω την ε, παραδοσία και την παρουσία του, Επιτροπου, του εισηγητή τη Επιτροπή ε, Προπολογισμού εδώ στην δική μα Επιτροπή και θα μιλήσω ρουμάνικα. Σας ευχαριστώ. Γιατί προφανώς θα πρέπει να τα συζητήσουμε αυτά πριν ε, ξεκινήσει η δημοσιονομική διαδικασία. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και όλες αυτές τις ε, πολιτικές σε ό,τι αφορά την τομέα των εξωτερικών υποθέσεων και θα ήθελα να καλωσορίσω την πρόσφατη ε, έγκριση των κατευθυντηρίων γραμμών για τον προεπιλογισμό του 2018 που αναφέρει και τα θέματα εξωτερικής πολιτικής τα οποία θα πραγματευτεί η Επιτροπή μας και θα βεβαιωθούμε ότι θα αποτυπώνονται στον προπολογισμό του επόμενου έτους και ο κύριος Μόρεσαν ήδη ανέφερε κάποια από τα θέματα αυτά. Αυτές οι προτεραιότητες λοιπόν περιλαμβάνουν ε, συνεχιζόμενη δημοσιονομική υποστήριξη από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ε, κρίση του προσφυγική, ε, χρηματοδότηση διευκολύνσεων για τους πρόσφυγες όπως αυτή της Τουρκίας και χρηματοδότηση των βαθύτερων αιτιών της προσφυγικής κρίσης. Αυτό δεν θα πρέπει να έχει αρνητικό αντίκτυπο, ωστόσο για τη χρηματοδότηση πολιτικών και εργαλείων ε, άλλων που εμπίπτουν στην ε, πολιτική εξωτερικών υποθέσεων. Θα πρέπει ο προπολογισμό να είναι επαρκή για να έχουμε και ένα κύρο στι δράσει μα και να μπορούμε να έχουμε και ένα αντίκτυπο, σε ό,τι αφορά τα μέσα που χρησιμοποιούμε το ΕΛΚ και οι υπόλοιπε πολιτικές ομάδες πάντα ήταν υπέρ αυτού του μέτρου. Ύστερα, έχουμε άλλα τέσσερα μέτρα και ζητήματα τα οποία σημαντικό είναι να τονιστούν. Και ως εισηγητής για τη γνωμοδότηση αυτή, της γνωμοδότησης αυτής στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, θα εξετάσουμε προσοχή τις προτάσεις ε, του Συμβουλίου. Σε ό,τι αφορά τους τέσσερις αυτούς τομείς, λοιπόν. Καταρχάς, πολιτική διεύρυνση και υποστήριξη των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Πολλές χώρες ε, στην περιοχή αυτή είναι εν δυνάμει υποψήφιες χώρες ή υποψήφιες χώρες και σήμερα αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες σε ό,τι αφορά θέματα δημοκρατίας, εντάσεις και τριβές που ανακύπτουν Μακεδονία, Αλβανία, Κοσφοπέδιο, Αυτά παρατηρούνται παντού, ακόμα και στο Μαύρο Βούνιο. Φυσικά υπάρχει και το θέμα του ΝΑΤΟ, υπάρχει και η Βοσνία, είμαι και συγκεκριτή για τη χώρα αυτή και ανακύπτουν λοιπόν τριβέ στι χώρε αυτέ και δεδομένων όλων αυτών θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στην καλή διακυβέρνηση, υποστηρίξη τη καλή διακυβέρνηση ε, στι χώρε αυτέ και να υποστηρίξουμε ασφαλώ και την καταπολέμηση τη διαφθόρα. Παράν τούτου. Νομίζω ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε την βελτίωση της δημόσιας διοίκησης, ανεξαρτησίας του τύπου, ρόλο της κοινωνίας πολιτών. Όλα αυτά είναι σημαντικά να αναφέρονται και νομίζω ότι οι στόχοι αυτοί μπορούν επίσης να επιτευχθούν και να αναφέρονται ασφαλώς σε ό,τι αφορά και την Τουρκία. Έγινε χθε η συζήτηση για την Τουρκία, παρουσιάστηκε και η έκθεση της Κατυπήρη για την ε, έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα πρέπει να επανοριστεί ενδεχομένω η σχέση μα με την Τουρκία, αλλά οι στόχοι αυτοί, η καταπολέμηση, τη διαφθορά και το καταξή, νομίζω ότι μπορούν επίση να εφαρμοστούν και σε διαφορά την Τουρκία, όπω και στα Δυτικά Βαλκάνια. Κατά δεύτερον, η υποστήριξη των ε, γειτονικών χωρών και κυρίω ε, των χωρών τη ε, Ανατολική Γειτονία και τη Νότια Γειτονία. Η πολιτική γειτονίας ο στόχος έχει να διατηρηθεί η σταθερότητα στις νότιες και ανατολικές περιοχές και προφανώς να προωθηθεί και η ανάπτυξη στις γειτονικές αυτές χώρες. Ασφαλώς η πολιτική γειτονία θα πρέπει να έχει πόρους τρίτων. Επαρκής χρηματοδότηση για εξωτερικές πολιτικές και πολιτικές για την κοινή ασφάλεια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό γιατί αυτός ο τομέας ε, της πολιτικής ουσιαστικά ως στόχο έχει την οικοδόμηση ειρήνης, τη σταθεροποίηση αλλά και την εξασφάλιση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο διεθνές προσκήνιο. Και συχνά σε ό,τι αφορά τις εξωτερικές πολιτικές διαπιστώνουμε πόσο σημαντικός είναι αυτός ο τομέας για τους εξωτερικούς εταίρους μας. Και ναι, ολοκληρώνω που ήταν πρόεδρε. Είναι σημαντικό λοιπόν ο προπολογισμό να αντικατοπτρίζει και να αποτυπώνει, αν θέλετε, και τις φιλοδοξίες μας. Τέλος, να αναφέρω τη σημασία του μέσου για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γενικώ πώς βλέπουμε ότι τακτικά είναι υπό επίθεση τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι αρχές της δημοκρατίας. Αυτό το παρατηρούμε όλο και πιο συχνά. Η καθολικότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το καθήκον μας να προασπιζόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις δημοκρατικές αρχές σε όλες τις χώρες είναι κάτι το οποίο προφανώς ε, ισχύει ακόμα και θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τον κύριο Μούρεσαν εκ νέου που είναι εδώ σήμερα και είμαι βέβαιος ότι θα είναι καλή συνεργασία από το θέμα. Τον Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. This item is called exchange of views. Ε, αυτό το θέμα φέρει το τίτλο «Ανταλλαγή απόψεων», αλλά έχουμε χρονική πίεση γιατί ήρθαν οι προσκεκλημένοι μας από το Κόσοβο. Έχω τέσσερις ομιλητές, Καλνιέτε, Γκάλα, ε, Γκίλ και Φλέκενστάιν, τους εξής πέντε. Έξι, γράψτε παρακαλώ, σημειώστε τα ονόματα. Ποιος άλλος θέλει το λόγο. Θα κλείσω τον κατάλογο. Έξι ομιλητέ έχουμε. Ζητώ συγγνώμη, αλλά θα πρέπει να το περιορίσουμε σε 1,5 λεπτό. Και ο κύριο Πέτρελ, έβδομο. Άλλο παρακαλώ, έχουμε χρόνο. Ο κύριο Επιτίδιο, 8. Ωραία. Έκλεισε ο κατάλογο. 1,5 λεπτό έκανε στου 8 ομιλητέ, γιατί μα περιμένουν οι ε, προσκεκλημένοι μα από το Κουσικοπέδιο. Thank you. Κύριε Γκέλ, ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και σαν Secret για την ανταλλαγή απόψεων. Είμαι σχεδόν συγκήτρια από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες και χαίρομαι που έχουμε την ευκαιρία αυτή να ανταλλάσσουμε απόψη. Και η συνεργασία των δύο επιτροπών μας σε προπολογισμού και εξωτερικό είναι πολύ σημαντική. Όπως και πέρσι, φαντάζομαι και φέτος εξωτερικές δράσεις ε, είναι πολλές και προκλήσεις της Ένωσης. Ήδη έχουμε συζητήσει τα θέματα, ε, να δούμε ποιε είναι οι αιτίε ε, των σειράξεων που σταθεροποιούν την περιοχή μας, στη γειτονία μας. Πρώτα το προσφυγικό, μετά η συνεργασία με τους εταίρους μας για την κλιματική αλλαγή και ενίσχυση των σχέσεων με στρατηγικούς εταίρους. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να πορευθούμε σε ταραγμένα νερά παγκόσμια. Ε, έχουμε πολλές προκλήσεις, πολλά προβλήματα και χρειάζεται και ο αντίστοιχο ε, προπολογισμό. Με ε, τη δέουσα ευελιξία, το μέσο ευελιξίας, ε, το αποθεματικό για τα κατεπήγοντα. Δεν έχει συμφωνηθεί ακόμα το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και το γνωρίζω αυτό, αλλά θα πρέπει να έχουμε κάποια ιδέα για τις οροφές, για τα όρια της αναθεώρησης. Όπως και πέρσι, εμείς ε, θα ε, ελέγχουμε πάρα πολύ και θα εκφράζουμε τον προβληματισμό μας για τα τα πιστευματικά ταμεία. Γιατί ε, ουσιαστικά μπορεί να καταλήξει αυτή η ιστορία στο να παίρνουμε από τον ένα χρήματα για να τα δίνουμε σε κάποιον άλλον. Ε, και ανησυχώ και για την Τουρκία, για τη χρηματοδότηση ε, του προσφυγικού και κάτι άλλο. Αν τελειώνω, όχι δεν μπορείτε να τελειώσετε. Το πρόγραμμα επενδύσεων που είναι πολύ σημαντικό για την ομάδα μας και έχει πολύ μεγάλη σημασία θέλουμε να εξαλείψουμε τη φτώχεια, να αντιμετωπίσουμε τη μετανάστευση και να υπάρχει προσθετικότητα αυτά και ε, συνοχή στην πολιτική. Ε, κοιτάξτε, έχουν έρθει άνθρωποι από το Κωσυφοπέδιο και περιμένουν απ' έξω. Από εσά θα εξαρτηθεί. Ε, παρακαλώ, η κυρία Καλνιέτη, τηρήστε το χρόνο σας να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Θα μπω αμέσω στο θέμα χωρίς να επενέσω τον εισηγητή. Ξέρει πόσο τον εκτιμώ και τον ίδιο και το έργο του. Στην έκθεση Φωτίγκα, εμεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τονίσαμε τη σημασία διεύρυνση ε, τη STATCOM στην υπηρεσία εξωτερική δράση από 8 μέλη δηλαδή να έχει 16 υπαλλήλου. Μέχρι τώρα δεν υπήρξε υποστήριξη του αιτήματο αυτού από τα κράτη-μέλη. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν το στήριξε στον προηγούμενο προπολογισμό. Και ρωτώ τον εισηγητή τώρα πώ διαφαίνονται τα πράγματα να εξελίσσονται ε, στον προπολογισμό. Θα έχουμε μεγαλύτερο ποσό για τη Στάτκομ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Σάντρα. Ο κύριος Φλέκενστάιν. Πάρα πολύ σύντομα και στα αγγλικά. Συμφωνώ πάρα πολύ με τα όσα είπε ο φίλος Πρέντα. Θα πρέπει με την ησυχία μας να μελετήσουμε σε βάθος τα θέματα αυτά. Δώσατε πολλά παραδείγματα ε, που πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα για να ασκούμε καλύτερη πολιτική. Έχω μια ερώτηση προς Γιατί δεν το κατάλαβα κύριε αν Στο τέλος της παρουσίασης μίλησατε για διάφορα έργα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει το Α ή το Β και εμείς λέμε, προτιμούμε το Α. Ή καλύτερα να έχουμε τις δικές μας ιδέες και να μην είμαστε παρακολούθημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Α, Β ή Γ. Εμείς είμαστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σολέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και... Πάρα πολύ σύντομα. Θα πρέπει να έχουμε τους πόρους για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το να έχει μια σταθερή γειτονία. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν απαιτεί μόνο πολιτικές ικανότητες και πολιτική βούληση, αλλά απαιτεί και πιστώσεις. Το θέμα δεν είναι μόνο να σταματήσουμε τους πρόσφυγες να έρχονται στην Ευρώπη, απαιτεί, αυτό είναι κάτι που θέλει μια άλλη συζήτηση, αλλά να προωθήσουμε γενικότερα τη δικαιοσύνη και την δημοκρατία στις γειτονικές χώρες. Απαιτούνται χρήματα λοιπόν και για το μέσο εταιρικότητας, όπως επίσης και για το μέσο σταθερότητας και ειρήνευσης. Και να υπογραμμίσω επίσης ότι δεν συμφωνούμε στον ενθουσιασμό τον οποίο εκφράσατε όταν μιλήσατε για τις αμυντικές πολιτικές και την έρευνα στον τομέα της άμυνας. Γκάλερ. Σας ευχαριστώ και την συντομία. Υποστηρίζω αυτά που είπε και η κυρία Καλνιέτε για τα πλατικά προγράμματα απόλυτη υποστήριξη και χαίρομαι ιδιαίτερος που το έθιξες το θέμα της έρευνας για την άμυνα ότι θα πρέπει να το δούμε πιο μακροπρόθεσμα το θέμα αυτό και στην επόμενη δημοσιονομική περίοδο και να δώσουμε αυτή την ε, μακροπρόθεσμη διάσταση. Από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό θα προταθεί αυτόματα, αλλά και από πλευρά μα θα θέλαμε να πούμε ότι δεν πρόκειται να βάλουμε προσκόμματα και εμπόδια προ την όλη αυτή τη διαδικασία. Ευχαριστούμε πολύ. Θα σα ευχαριστούμε κύριε Γκάλερ και τέλο ο κύριο Πέτερλε. Ε, το έθεσαν το ερώτημα που θέλω να θέσω, οπότε δεν χρειάζεται να μιλήσω. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μούρεσαν θα ήθελε να πάρει το λόγο για να απαντήσει. Εν συντομία, εν συντομία, Πρόεδρε, επειδή περιμένουν έξω και οι μας σε ό,τι αφορά τι ε, τις αιτίε τη της ε, μετανάστευση. Είναι ακριβώ. Ο κόσμο φεύγει γιατί δεν έχει εκπαίδευση, υποδομέ, ε, τρόφιμα, νερό, δεν έχει ασφάλεια και το καθεξή. Προφανώ, προφανώ όλα αυτά θέλουμε να τα πετύχουμε και αυτά προσπαθούμε να στοχεύσουμε σε ό,τι αφορά και τη γειτονία, την πολιτική γειτονία προς την ε, Τρονοτό. Κατά δεύτερον, το είπε και ο κύριος ε, Πρέντα σε ό,τι αφορά τα θέματα ε, πολιτικής ε, Άμυνα και εξωτερική πολιτική, Αυτό δεν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σε ό,τι αφορά και το πολιτικό δημοσιονομικό πλαίσιο. Και εδώ πέρα θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη. Υποστηρίζουμε λοιπόν από πλευρά μου και την ιδέα αυτή και τε, ύστερα αναφέρθηκα και στην πολιτική γειτονία προ Ανατολά και προ την Νότο. ο κ. Πρέντα αναφέρεται στα Βαλκάνια. Αλλά θα έπρεπε να είμαστε έτοιμοι. Γιατί αν υπάρχουν εξελίξει εκεί στην Αλβανία, στην ε, πρώην Ιεκοσλαβική Δημοκρατία τη Μακεδονία, στη Βοσνία, αν υπάρξουν εκεί εξελίξει και αν οι εξελιξει ε, απαιτήσουν να κάνουμε κάτι παραπάνω για την καταπολέμηση τη διαφθορά την πράσινη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να δράσουμε. Και το λέω αυτό και προ την κυρία Καλνιέτε. Ε, κατέθεσα ένα πολιτικό πρόγραμμα για να υπάρξει ο προπολογισμό και αύξηση του προπολογισμού με 3 εκατομμύρια ευρώ για του χρόνου για όλα τα πολιτικά προγράμματα για να υπάρχει μια ελεύθερη αξιολόγηση για να δούμε κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δώσει την ανάλογη πρικοδότηση. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν τι θα ζητήσουμε και εμείς επιπλέον σε ό,τι αφορά τις δημοσιονομικές ε, τροποποίησεις στο φθινόπωρο. Να δούμε τι θα καταθέσει λοιπόν ως πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο σχέδιο προπολογισμού και μετά είμαστε έτοιμοι να αυξήσουμε και τον προπολογισμό του, του Stratcom. Γιατί ε, αν δεν υπάρχει μακροπρόθεσμη σταθερότητα σε ό,τι αφορά το προσωπικό. Αν κατά δεύτερον, ε, το η χρηματοδότηση της είναι περιορισμένη. Τι σημαίνει αυτό, ότι μπορούν να κάνουν και κάποια πράγματα σε ό,τι την εποπτεία, αλλά όχι και κάτι για να καταπολεμήσουν ενεργά την προπαγάνδα. Κατά δεύτερον, βασίζονται σε ένα δικτύο εθελοντών. Όλα αυτά λοιπόν είναι πολύ στον αέρα. Χόκα. Από κάποιε χώρε λαμβάνουν πληροφορίε, από κάποιε άλλε δεν λαμβάνουν επαρκέ πληροφορίε και όσοι συμβάλλουν τελικά είναι δημοσιογράφοι από μικρέ ΜΚΟ για την, η δουλειά τους για τη Stratcom είναι να επιβαρύνει ουσιαστικά την οργάνωσή τους. Δηλαδή τους ε, στερεί χρόνο από τις καθημερινές τους εργασίες. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν πώς η Stratcom μπορεί να μπει σε μια σταθερή, στεναρή μακροπροθεσμή βάση. Αλλά καταρχάς πλωτικά προγράμματα και κατά δεύτερον επιπρόσθετες τροποποιήσεις στον προπολογισμό εφόσον και αν χρειαστούν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Μάλιστα, λέει και ο Πρόεδρος. Ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ζίγκριτ Μούρισαν για την ανταλλαγή αυτή απόψεων για τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2018. Ελπίζω ότι η οι παρεμβάσει των συναδέλφων ήταν χρήσιμε για τη μελλοντική σα εργασία. Θα συνεχίσουμε την καλή συνεργασία, προφανώ. Και τώρα, 10 και 37 είναι η ώρα. Μπορούμε να ε, υποδεχτούμε του προσκεκλημένου μα από το 20 Μα μόλι μου είπατε ότι ήταν έξω και περίμεναν. Μα πείτε του να μπουν μέσα, αν θέλετε. Ladies and gentlemen, dear colleagues, we come to... Αγαπητοί συνάδελφοι, περνάμε στο 17. Ανταλλαγή απόψεων με τον Υπουργό Εξωτερικών του Κωσυφοπεδίου, τον Ένβερ Χότζα. Έχουμε μία ώρα για αυτήν την ανταλλαγή απόψεων Γύρω στις 11.30 θα περάσουμε στο επόμενο θέμα. Να καλωσορίσω τον κύριο Υπουργό για μια ακόμη φορά στην Επιτροπή μας. Έρχεστε συχνά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είστε κάποιος με τον οποίο θέλουμε να επικοινωνούμε. Συνοδεύεστε από τον πρέσβη του Κοτσιφοπεδίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ήθελα επίσης να καλωσορίσω δύο συναδέλφους από το Κοινοβούλιο του Κοσφοπεδίου. Έχουμε την πρόεδρο της Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, την κυρία Έμινη, και να καλωσορίσω επίσης και τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων στην Πρίστινα, τον κύριο Έλμι Ρέτσιτσα. Ελπίζω να τα είπα σωστά. Τους καλωσορίζω και αυτούς. Ο κύριος Χότζα είχε μιλήσει ξανά εδώ στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη σταθεροποίηση που έγινε στις 20 και στις 21 Απριλίου ε, και ο Πρωθυπουργός Μουσταφά ήταν την προηγούμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες. Για μια ακόμη φορά λοιπόν σας καλωσορίζουμε και θα σας δώσω το λόγο έτσι ώστε να αναφερθείτε σε όλα τα θέματα τα οποία παρουσιάζουν σημασία για την χώρα σας, την κυβέρνησή σας. Είμαι σίγουρος ότι θέλετε να αναφερθείτε και στα τελικά βήματα για την απελευθέρωση των θεωρήσεων, όπως επίσης ε, και την ε, συμφωνία ε, για τον καθορισμό σύνορων με το Μαυροβούνιο, για την ενίσχυση του κράτους δικαίου, την καταπολέμηση της διαφθοράς κτλ. κτλ, κτλ. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και το φίλο David. Αγαπητά μέλη του Κοινοβουλίου, αγαπητά μέλη του Κοσφοπεδίου και της περιοχής, σας είμαι ευγνώμων για την πρόσκλησή σας για να δούμε το πώς έχει η κατάσταση στη χώρα μου και γενικότερα στην περιοχή. Να ξεκινήσω ευχαριστώντας σας για μια ακόμη φορά για την σοβαρή στήριξη την οποία μας παρέχεται τα τις τελευταίες δύο δεκαετίες σας ευχαριστούμε που μας υποστηρίζετε στην πορεία για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, όπως επίσης μας υποστηρίζετε έτσι ώστε να γίνουμε πλήρες μέλος της διεθνούς κοινότητας και της διεθνούς κοινωνίας. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να υπάρξει πρόοδο στο κοσφοπέδιο αν δεν είχαμε τη δική σας υποστήριξη. Παρακολουθούμε πολύ κοντά όλες τις συζητήσεις τις οποίες έχετε συχνά στα κοινοβούλια σας και σας ευχαριστώ για τα πρόσφατα ψηφίσματά σας ε, γύρω από την κατάσταση στη χώρα μου. Και οι συστάσεις σας για μας σαν κυβέρνηση είναι βασική αναφορά για την καθημερινή μας απασχόληση. Σήμερα είναι μια σοβαρή, θα έλεγα, στιγμή για την, ε, με την υποστήριξη της κυρίας Λούνατσεκ, φίλης του Κοσφοπεδίου, ξεκινήσαμε την ομάδα φίλων ε, του Κωσυφοπεδίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι ένα πρώτο σημαντικό νομίζω βήμα για το Κωσυφοπέδιο. Είναι μια διαδικασία βραχυπρόθεσμη αλλά και μακροπρόθεσμη που θα μας επιτρέψει να ανταλλάσσουμε απόψη με μέλη των, του Κοινοβουλίου σας. Σαν μέλος της ε, κυβέρνησης εμείς ε, εκτιμούμε ιδιαίτερα το θεσμικό αυτό όργανο και εκτιμούμε την υποστήριξή σας σε όλα τα επίπεδα. Αυτό το οποίο θα ήθελα είναι να έχουμε λοιπόν μια σωστή διαδικασία ερωτήσεων-απαντήσεων. Εγώ είμαι Βαλκάνιος πολιτικός και μερικές φορές θέλουμε μια ώρα για να πούμε αυτά τα οποία έχουμε να πούμε και θα χρειαζόμουν, μια και είμαι και καθηγητής, ε, δύο ώρες για να σας περιγράψω σωστά την κατάσταση ε, στο Κοσφοπέδιο και τα Βαλκάνια. Δεν θα το κάνω όμως αυτό. Θα προσπαθήσω να σας ενημερώσω για τα βασικά θέματα τα οποία έχουμε μπροστά μας και ελπίζω να ακολουθήσει η συζήτηση. Εξελέγει τέσσερις φορές ε, μέλος του Κοινοβουλίου στο Κοσφοπέδιο και ξέρω πόσο σημαντικό είναι να είσαι μέλος ενός τέτοιου οργάνου. Ε, το πώς πρέπει να δει κανείς το κοσφοπέδιο το 2017, τι είναι το κοσφοπέδιο. Εμείς προετοιμάζουμε το κοσφοπέδιο που είναι η νεότερη ε, χώρα και το νεότερο κράτος των Βαλκανίων και της Ευρώπης φυσικά <clears throat> για τις σχέσεις με την γειτονία. Έχουμε θα έλεγα μια σταθερή πολιτική σχέση με την γειτονία μας Αν θέλουμε να περιγράψουμε το κοσφοπέδιο με απλούς όρους θα πούμε σταθερότητα, ασφάλεια και προβλεψιμότητα. Νομίζω ότι αυτά τα τρία χαρακτηριστικά είναι σημαντικά για να καταλάβει κανείς το τι έχουμε πετύχει μέχρι τώρα. Έχουμε μια περιοχή και μια γειτονία η οποία αμφισβητείται εσωτερικά, ε, δεν έχουμε σε πολλές χώρες της περιοχής εσωτερικές καταστάσεις σταθεροποιημένες και έχουμε επίσης και ε, πολλούς παράγοντες τα τελευταία χρόνια, ξένους προς την περιοχή, που είναι δραστήριοι τα τελευταία τρία χρόνια. Ε, what Αυτό το οποίο θέλω να πω years of είναι ότι μετά από 10 χρόνια ανεξαρτησίας το κοσυφοπέδιο είναι το λεγόμενο success story της περιοχής. Πετύχαμε εμείς να χτίσουμε το κράτος μας από το μηδέν και αν δεν είχαμε τη δική σας υποστήριξη δεν θα το πετυχαίναμε. Δεν έχουμε μόνο την πιο σταθερό πολιτικό τοπίο, έχουμε επίσης και μια εισοδηματική και μακροοικονομική σταθερότητα, τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη του ΑΕΠ 4 με 4,5% ήταν κατέτος πολύ σημαντική. Πέραν της ενίσχυσης των κρατικών δομών, που ήταν ο βασικός στόχος της κυβέρνησής μας τα τελευταία χρόνια, Δεύτερος στόχος ήταν η διεθνής ενίσχυση της παρουσίας του κοσφοπεδίου. Μας έχουν αναγνωρίσει μέχρι τώρα 140 χώρες 114 λέει ο κύριος Χόρζαϊ. Και θα ήθελα να επαναλάβω για μια ακόμη φορά ότι υπάρχουν πέντε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ακόμα δεν έχουν αναγνωρίσει το παιδιό να πάρουν την απόφαση να το κάνουν. Είναι ένα πολιτικό εμπασί περιπτώσει γεγονός, εμείς έτσι κι αλλιώς θα μείνουμε και είμαστε και θα μείνουμε ανεξάρτητο κράτος και γι' αυτό πρέπει να μας αναγνωρίσετε και αυτό θα κάνει και την Ένωση και τη χώρα μας ισχυρότερη. Εγώ παρακολούθησα τις διαδικασίες διαπραγμάτευσης το 2006 και το 2007 που οδήγησαν σε ανεξαρτησία τη χώρα μου. Ήταν μια διαδικασία λοιπόν η οποία δεν μου έδινε τότε την δυνατότητα να σκεφτώ ότι μετά από 10 χρόνια ότι θα ερχόμουν εδώ και θα υπάρχουν πέντε χώρες που δεν μας έχουν ακόμα αναγνωρίσει. Ζητώ την υποστήριξή σας λοιπόν και ζητώ την υποστήριξη των πέντε κυβερνήσεων για να πάρουν αυτή τη σημαντική απόφαση για μας. Σχετικά τώρα με τη συμμετοχή του κοσφοπεδίου στη διεθνή κοινωνία και τη διεθνή κοινότητα, ε, μέχρι τώρα έχουμε γίνει μέλη σε 50 περιφερειακές, ευρωπαϊκές και διεθνείς οργανώσεις. Εδώ και λίγες εβδομάδες ε, γίναμε μέλη της Διεθνούς Οργάνωσης Τελωνιακών Αρχών ε, που μετά από το Δέλτα Νιτάφ και την Παγκόσμια Τράπεζα ε, είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό για μας στον τομέα των τελωνιακών διαδικασιών. Επίσης στην UNESCO, στην Interpol και νομίζω ότι η υποστήριξή σας επιδιώκουμε να μπούμε και θα είναι σημαντική. Η πιο σημαντική μας σχέση όμως είναι με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είστε ο πιο σημαντικός μας εταίρος. Είμαι θα ευγνώμονες λοιπόν που μας υποστηρίζετε για να υπογράψουμε ε, μια συμφωνία σταθεροποίησης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και ως πολιτικός θα ήθελα να πω ότι δεν είναι μόνο κάτι το πάρα πολύ σημαντικό αλλά και ταυτόχρονα εσωτερικά θα έλεγα είναι το καλύτερο πλαίσιο για τον εξυγχρονισμό της πολιτικής μας, της κοινωνίας μας, της οικονομίας μας και νομίζω ε, είναι κάτι το οποίο χρειάζεται στα Βαλκάνια όχι μόνο τα τελευταία 10-20 χρόνια αλλά τα τελευταία 200 χρόνια. Is beyond Europe, the region has another speed. Εμείς λοιπόν λειτουργήσαμε σε διαφορετική ταχύτητα από την υπόλοιπη Ευρώπη και θα πρέπει να ενταχθούμε στις διαδικασίες εξυγχρονισμού ε, κάτι το οποίο δεν έγινε τα τελευταία 200 χρόνια για τη χώρα μου. Τον προηγούμενο Δεκέμβριο είχαμε το πρώτο Συμβούλιο Σταθεροποίησης Ευρωπαϊκής Ένωσης με την κυβέρνηση του Κοσφοπεδίου. Παρέστη η Μογκερίνη και ο Μουστάφα, ο Πρωθυπουργός, πριν λίγες μέρες συνεδρίασε και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή, η Διακοινοβουλευτική. Πολλοί φίλοι που είναι εδώ τώρα ήταν στην Πρίστινα και τους ενημερώσαμε για το τι έχουμε πετύχει μέχρι τώρα. Το πιο σημαντικό θέμα το οποίο έχουμε εσωτερικά είναι η εφαρμογή της Συμφωνίας Σταθεροποίησης, όπως επίσης και η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Ατζέντας για μεταρρυθμίσεις. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να τα ολοκληρώσουμε όλα αυτά τα επόμενα δύο χρόνια. Και όταν μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτή την φάση, τότε το κοσφοπέδιο θα ζητήσει ένα διαφορετικό καθεστώς, γιατί είμαστε η μόνη χώρα που δεν είμαστε υποψηφία χώρα στην περιφέρεια και θέλουμε την υποστήριξή σας. Το Κοσφοπέδιο λοιπόν προς το παρόν είναι η μοναδική χώρα η οποία δεν έχει την δυνατότητα καθεστώτος απελευθέρωσης των θεωρήσεων και γι' αυτό θέλουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε σαν κυβέρνηση για να καλύψουμε όλα τα κριτήρια τα οποία και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται και τις επόμενες εβδομάδες θα έχουμε σημαντικές αποφάσεις του Κοινοβουλίου για την επικύρωση της ε, συμφωνίας της συνοριακής με το Μαυροβούνιο. Και ελπίζω και γι' αυτό να τύχουμε της δική σας υποστήριξης και της υποστήριξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έτσι ώστε να μπορούν να ταξιδεύουν χωρίς θεωρήσεις οι πολίτες του κοσφοπεδίου. Είμαστε μια ζωηρή, η πιο ζωηρή κοινωνία, η νεότερη ηλικιακά κοινωνία στα Βαλκάνια, και το να παραμένει το Κοσφοπέδιο σαν ένα απομονωμένο νησί δεν είναι προς όφελος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πόσο μάλλον υπέρ των συμφερόντων των πολιτών μας. Να σας ενημερώσω επίσης ότι τα τελευταία 5-6 χρόνια όχι μόνο συνεχίσαμε τον διάλογο με τη Σερβία, αλλά νομίζω ξεκινήσαμε να οικοδομούμε μια νέα σχέση με τις δύο χώρες. Δεν λέω ότι οι σχέσεις έχουν αλλάξει πραγματικά, αλλά σίγουρα έχουν βελτιωθεί. Μπορέσαμε να υπογράψουμε 20 συμφωνίες και η βασική προτεραιότητα για μας είναι το πώς ε, θα εφαρμοστούν όλες οι συμφωνίες οι οποίες έχουμε πετύχει μέχρι τώρα, όπως την ενέργεια, την δικαιοσύνη, και της, ε, ε της Ενώσης των Δήμων και Κοινοτήτων, των κοινοτήτων βασικά, είναι στόχος μας ε, για τους επόμενους μήνες. Ο διάλογος αυτός έχει αλλάξει κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό θα έλεγα, θα πρέπει να το δείτε σε ευρύ ιστορικό πλαίσιο. Η σχέση κοσυφοπεδίου Σερβίας ήταν πάντα αυτό που ονομάζουμε zero sum game, δηλαδή πάντα κάποιος χάνει για να κερδίσει ο άλλος. Έχει αλλάξει τώρα η φύση της σχέσης μας, δεν ισχύει αυτό και εμείς σαν κυβέρνηση πιστεύουμε ότι ο διάλογος αυτός θα πρέπει να έχει ξεκάθαρους στόχους και ένας από τους πιο σημαντικούς στόχους του διαλόγου αυτού είναι η αμοιβαία αναγνώριση. Νομίζω ότι χωρίς αυτό ο διάλογος ανάμεσα στις δύο χώρες θα είναι τελικά άχρηστος και κενός νοήματος. Η αμοιβαία αναγνώριση θα πρέπει να είναι ο στόχος τον οποίο θα έχουμε ε, σαν στρατηγική για τα επόμενα χρόνια. Βρισκόμαστε λοιπόν σε διάλογο με την Σερβία, όχι μόνο για να βελτιώσουμε τις σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες, αλλά γιατί κατανοούμε περιφερειακά τη σημασία που έχει ένας τέτοιος διάλογος για όλη την περιοχή πέραν των σχέσεων Κοσφοπεδίου Σερβίας έχουμε και άλλες δύο ιστορικές προκλήσεις οι οποίες δεν έχουν αντιμετωπιστεί ακόμα. Η μία από αυτές είναι το θέμα του ονόματος της Μακεδονίας, λέει ο κ. υπουργό. Δεν θα ασχοληθώ ιδιαίτερα με αυτό, δεν είναι κάτι το οποίο ανήκει στις αρμοδιότητές μου, αλλά θα θέλαμε η περιφέρεια να προχωρήσει. Και δεύτερον έχουμε την εσωτερική κατάσταση στη Βοσνία, η οποία μας ανησυχεί ιδιαίτερα. Γιατί αν η χώρα αυτή ε, καταρρεύσει, τότε θα έλεγα θα κινδυνεύσει όλη η περιοχή. Εμείς προσπαθούμε λοιπόν να προωθήσουμε τις περιεφηριακές πολιτικές, οι χώρες να βοηθούν η μία την άλλη και όχι να αποκλείουν η μία την άλλη ο πολιτικός διάλογος τον οποίο είχαμε μέχρι τώρα σε επίπεδο πρωθυπουργών και, και προέδρων συνεχίζεται και θα πρέπει νομίζω όλες οι χώρες να συμμετέχουν. Θα βοηθήσει και σε επίπεδο αντίληψης ανάμεσα σε κυβερνήσεις, ανάμεσα σε αρχές, ανάμεσα σε πανεπιστημιακά ιδρύματα κτλ. Κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι η υποστήριξη του εκλεκτού σας σώματος, η υποστήριξη των ευρωπαϊκών οργάνων και της Ένωσης γενικότερα έχει οδηγήσει σε αλλαγές στην περιφέρειά μας τα τελευταία 20 χρόνια. Η μισή περιοχή μας ανήκει στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και το άλλο μισό είναι σε διαφορετικές φάσεις πορείας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντως θεωρούμε ότι τα τελευταία δύο-τρία χρόνια λόγω ακριβώς κάποιων ιστορικών προκλήσεων οι οποίες δεν έχουν ακόμα αντιμετωπιστεί όπως οι σχέσεις Σερβίας, τα η Βοσνία κτλ. κτλ. Υπάρχει ένας μακρύς κατάλογος θεμάτων όπως τα μειονοτικά θέματα, τα θέματα του καθορισμού συνόρων. It's, um, η κατάσταση λοιπόν αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ανοιχτή εκκρεμότητα θα έλεγα. Όταν ήμουν εδώ πριν 3-4 χρόνια, το 2013 νομίζω που είχα έρθει εδώ να πάρω το λόγο, εκείνη την εποχή ήμουνα λίγο πιο θετικός για την περιοχή γιατί ήταν το 2014 σημαντικό έτος ε, ενετάχθη η Κροατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπήρξαν θετικές αλλαγές και τον Απρίλιο του 2013 το Κωσυφοπέδιο και η Σερβία κατέληξαν σε μια ιστορική συμφωνία. Ήταν λοιπόν μια πολύ καλή χρονιά το 2014. Δεν μπορώ όμως δυστυχώς να πω ότι θα μπορούσα να θεωρήσω το ίδιο για το τι συμβαίνει φέτος. Δεν είναι τόσο ελπιδοφόρα η κατάσταση. Θα ήθελα λοιπόν να προσπαθήσετε να αυξήσετε την προσοχή σας προς την περιοχή μας, να στηρίξετε τις διαδικασίες που ξεκίνησαν πριν 20 χρόνια και νομίζω ότι με την υποστήριξή σας θα πετύχουμε κάτι καλύτερο στο μέλλον. Ε, σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας και θα ήθελα να έχω μια ειλικρινή συζήτηση ε, μαζί σας, όσο ειλικρινής μπορεί να είναι ένας υπουργό εξωτερικών βέβαια. Ευχαριστώ. Ένβερ, για τα σχόλιά σας, τα εισαγωγικά και τις παρατηρήσεις σας. Πόσο ομιλητές έχουμε? 11 παρακαλώ συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο. Επειδή θέλουμε να ακούσουμε και την απάντηση του κυρίου Χότζαη, θα πρότεινα δύο λεπτά για κάθε ομιλητή. Αρχίζουμε. Η κυρία Λούνατσεκ πρώτη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε, κύριε Υπουργέ, στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Θα ήθελα να επαναλάβω και αυτό που είπατε και εσείς σήμερα το πρωί Πολλά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήρθαν, 11 μέτρησα εγώ και κάποιοι άλλοι δεν μπόρεσαν να έρθουν και το γνωρίζω αυτό ε, στην ε, εγγενία, στα εγγένεια της ομάδας ε, φιλίας Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Κοσυφοπεδίου και δύο εξέχοντα μέλη της Βουλής σας Πρόεδρος Επιτροπής Εξωτερικών και Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης και εσείς ο ίδιος. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και σας καλωσορίζω. Ήταν πολύ καλή η συνεδρίαση και ε, ήταν σκόπιμο να έχουμε πιο συχνά τέτοιες ανταλλαγές γιατί βοηθάει στην αμοιβαία κατανόηση για κάποια κρίσιμα ζητήματα που παραμένουν ή που θέλουμε να ε, μάθουμε. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ορισμένα από τα θέματα που θέσατε και θα προσπαθήσω να τηρήσω και το δίλεπτο μου. Θα περιστώ σε δύο. Στην ε, απελευθέρωση θεώρησης διαβατηρίων και την κατάσταση στην περιοχή. Τα έχουμε ξανασυζητήσει αυτά τα θέματα της Βίζας επανειλημμένως. Θα πρέπει ε, η Βουλή σας να ε, ψηφίσει για το θέμα των συνόρων με το Μαυροβούνιο. Το ξέρω ότι δεν είστε μέλος Βουλής, αλλά είναι η τελευταία χώρα στην περιοχή που δεν μπορούν να ταξιδεύουν ελεύθερα οι πολίτες. Έχουμε μεγαλύτερες χώρες όπως είναι η Ουκρανία και η Γεωργία που δεν είναι στη διαδικασία διεύρυνσης, όπου έχει επέλθει η απελευθέρωση των θεωρήσεων και θέλω το συντομότερο να γίνει αυτό και για το κοσμοπέδιο και ξέρω ότι και η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου. Ε, θα πρέπει επιτέλους να προχωρήσετε στον ορισμό των οριστικών συνόρων με το Μαυροβούνι. Δεύτερον, πολύ σωστά είπατε ότι ε, παραμένουν ε, κάποια κράτη-μέλη, πέντε τον αριθμό που δεν έχουν αναγνωρίσει το κόσο υφοπαίδιο. Περίπου τα μισά και παραπάνω κράτη-μέλη των Ηνωμένων Εθνών σας έχουν αναγνωρίσει και θέλουμε να είστε μέλη του ΟΗΕ. Αλλά ε, επειδή αναφερθήκατε στην κατάσταση στην περιοχή, το έχουμε συζητήσει και εδώ στο Κοινοβούλιο και συμφωνώ μαζί σας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάπως απούσα από την περιοχή. Έχει χάσει την έγλη που είχε και φταίμε και εμείς γι' αυτό. Ε, δώστε μου μισό λεπτάκι. Είμαι εισηγήτρια για το Κόσοβο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, ξέρετε πόσο αυστηροί είσαστε εσείς όταν προεδρεύετε στην Ολομέλεια. Ε, λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά όχι, δεν μπορείτε να τελειώσετε. Οι κανόνε ισχύουν προ όλου, ακόμα και προ αντιπροέδρου. Εδώ μιλώ ω εισηγήτρια για το Κοσμοπέδιο, όχι αντιπρόεδρο. Μια πρόταση παρακαλώ να πείτε κυρία Αντιπρόεδρε. Η, επιτρο... η επιρροή ε, στην περιοχή της Ρωσίας και της Τουρκίας αυξάνεται και θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας και θα πρέπει να ενισχύσουμε την παρουσίαση, της, ε- της, παρουσίαση, συγγνώμη, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στο Κωσυβοπαίδιο και αλλού στην περιοχή και να μην τα αφήσουμε ως έχουν. Ευχαριστώ κυρία Λούνατσεκ. Στην Ολομέλεια να μου δώσετε ένα λεπτάκι παραπάνω, στο Στρασβούργο ραντεβού, σίγουρα. Λοιπόν, Έλκα. Ο κύριος Αντάκτουσον για δύο λεπτά το πολύ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ Εξωτερικών, χαίρομαι ε, που σας βλέπω στις Βρυξέλλες. Συναντηθήκαμε πριν από μισή ώρα με την αντιπροσωπή στην έναρξη των εργασιών της Ομάδας Φιλίας Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, Κόσυφο Παιδίου. Σας καλωσορίζω και εγώ στις Βρυξέλλες και στην Επιτροπή μας. Είχαμε εξαιρετική ανταλλαγή απόψεων στην Μικτή Κοινοβουλευτική πριν από μία εβδομάδα, κάτι τέτοιο στην Πρίστινα. Πολύ σημαντική συνεδρίαση με ανταλλαγή απόψεων για όλα τα μεγάλα θέματα που απομένουν να λυθούν σε ό,τι αφορά τη σχέση μας και την περαιτέρω ολοκλήρωση Είχα κάνει μια ερώτηση και στην Πρίστιν, μάλλον σήμερα το πρωί, και δεν απαντήθηκε για λόγους ε, χρονικούς. Και θέλω να το ξαναθέσω. Τι γίνεται με τη διαφθορά. Η διαφθορά είναι ένα από τα δύο εναπομείναντα ε, προαπαιτούμενα και επειδή επισκέφτηκα πολύ πρόσφατα τη χώρα σας, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Μάλλον το εξής δύο. Τι κάνετε για να διορθωθεί, για να αλλάξει η γενική αντίληψη στον κόσμο και στα μέσα ενημέρωσης που λένε ότι το μόνο ζήτημα που απομένει να λυθεί είναι το ζήτημα των συνόρων με το Μαυροβούνιο και πότε θα μπορέσετε να ασχοληθείτε με τα υπόλοιπα ε, όμως που έχουν να κάνουν με την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος. Θα με ενδιαφέρει να ακούσω την απόψή σας σχετικά. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ και τα ο κύριος Φρόιντ από τους Ζελιστές και Δημοκρατές. Ευχαριστώ πάρα πολύ πρόεδρε και θα ήθελα να συνεχίσω από εκεί που διακόψατε αγενέστατα την κυρία ε, Λούνατσεκ. Ο, αστείευομαι, αστείευομαι. Μα τι είναι, Αυστριακή αλληλεγγύη. Ε, ναι, ναι, ναι, η Αυστριακή φιλία πέρα από το πολιτικό φάσμα και τα πολιτικά μας προβλήματα, τα οποία ενδεχομένω έχουμε. Όχι. Θα ήθελα λοιπόν να συνεχίσω από εκεί που σταμάτησε η κυρία Λούνατσεκ. Έφερε τη ρωσική υπερβολή στην περιοχή και το έχουμε συζητήσει αυτό και στην ομάδα της φιλίας της περιοχής. Θα ήθελα να το θέσω αυτό όμως και να το ακούσω και την απάντησή σας σε αυτό το συγκείμενο. Ακούγονται φήμες και παραπάνω από φήμες ότι η Ρωσία προσπαθεί να παρέμβει στα Δυτικά Βαλκάνια. Να χρησιμοποιήσει, αν θέλετε, και να εκμεταλλευτεί την αδυναμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να προωθήσει τη δική της επιρροή στην περιοχή. Πείτε μας λοιπόν αυτό σε τι βαθμό παρατηρείται και στο Κωσυφοπέδιο. και σε τι βαθμό θεωρείτε ότι αυτό αποτελεί πρόβλημα για όλη την περιοχή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Επόμενος ομιλητή, ο κ. Νέατ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σα ρωτήσω για την εκρηκτική κατάσταση. Δεν θέλω να επιμείνω σε ερωτήσεις που έγιναν ήδη. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο που θεωρώ κεφαλαιόδου σημασία για την εκρηκτική κατάσταση στη Μακεδονία, λέει ο κ. Νάρτ, όπου οι γειτονικέ χώρε όμορες της Μακεδονίας, και μιλώ για την Αλβανία και το Κωσυφοπαίδιο, και φυσικά για την Ελλάδα και για τη Βουλγαρία, δεν κάνουν κάτι θετικό για να ηρεμήσουν τα πνεύματα εκεί που είναι εκρηκτική η κατάσταση. Έχουν προβλήματα οι δύο κοινότητες στη Μακεδονία. Η αλβανική κοινότητα και η άλλη που είναι επίσης τμήμα της Μακεδονίας. Για να λυθεί αυτό δεν χρειάζονται ομάδες αλληλεγγύης σε συνεργασία ε, του κοσφοπεδίου με τη Μακεδονία και την αλβανική κοινότητα συγκεκριμένα εννοώ. Ευχαριστώ κύριε Νάρτ. Και τώρα η κυρία Σουίτσα. Ευχαριστώ, David. Να ευχαριστήσω και τον Χωζαϊ που ήλθε σήμερα εδώ. Να σας συγχαρώ για την ομάδα φιλίας αυτή, την οποία και ξεκινήσατε σήμερα το πρωί. Στην οποία θα συμμετάσχω και εγώ. Γιατί θέλω να υποστηρίξω και την πρόοδο του κοσφοπεδίου. Αναφερθήκατε στην αρχή της παρέμβασής σας ότι σας προκαλούν, ε, αποτελούν πρόκληση κάποιοι μη ευρωπαϊκοί φορεί. Δεν τους κατανομάσατε, αλλά νομίζω ότι κατά νου έχετε τη Ρωσία, την Τουρκία. Δεν είπατε τίποτε για τις σχέσεις αυτές ε, Κωσυφοπέδιο-Τουρκία. Για διευκρινίστε παρακαλώ την σχέση αυτή. Επίσης, για μένα, ως αντιπρόεδρος της αποστολής αυτής για τη Βοσνία, Ζεγοβίνη και το Κωσυφοπέδιο, πρέπει να σας πω ότι η μοναδική πρόοδος η οποία διαφαίνεται είναι η συγχωγή του κώδικα, τηλεφωνικού κώδικα 038. Ε, 383, συγγνώμη. Ε, τι γίνεται, γιατί δεν μπορείτε να βρείτε συμφωνία για τα σύνορα με το Μαυροβούνιο μπορείτε να πείσετε το κοινοβουλίο σας, γιατί αυτό αποτελεί το μοναδικό εμπόδιο για σας για την απελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων. Μπορείτε να μας απαντήσετε γι' αυτό. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Η κυρία Βόρτα από τους Σοσιαλιστές και Δημοκρατές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πολύ χαίρομαι κι εγώ που έγινε σήμερα η εκκίνηση της Ομάδας Φιλίας Κοσφοπεδίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να πω δύο λόγια για κάποια από τα ζητήματα τα οποία θα πρέπει να ρυθμιστούν μετά τις συγκρούσεις ακόμα. Το κοσυφοπέδιο έχει νομοθεσία για τη συμπερίληψη των επιζώντων σεξουαλικής βίας και ε, συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία βετεράνων πολέμου και θυμάτων και αναφέρομαι στην νομοθεσία για τα δικαιώματα ε, των ε, θυμάτων, των αμάχων, των οικογενειών τους και το καθεξής. Οι πολιτική του κοσφοπεδίου επανειλημμένα έχουν υποσχεθεί να δώσουν υποστήριξη στις γυναίκες θύματα σεξουαλικής βίας, αλλά δεν έχει γίνει τίποτε προς το παρόν για την Πότε θα ξεκινήσει λοιπόν η Επιτροπή αυτή και τα ζητήματα αυτά να ρυθμίζονται στην πράξη και πότε οι επιζώντες αυτοί μπορούν να λάβουν πραγματικά βοήθεια από τον νόμο και να λάβουν συγκεκριμένα τη βοήθεια που χρειάζονται. Ε, εγώ και οι υπόλοιποι ευρωβουλευτές θα παρακολουθήσουμε πάρα πολύ στενά την υπόθεση αυτή μέχρι σότου να πραγματοποιηθούν αυτές οι υποσχέσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Βάιγκλ από τους ε, φιλελεύθερους από την Άλντα. Ο κύριος Ράντος, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον Υπουργό για τα εισαγωγικά του σχόλια. Πέρα από τα ζητήματα τα οποία αναφέρατε και τα οποία κυριαρχούν προφανώς το θέμα των σύνορων με το Μαυροβούνιο, το θέμα της καταπολέμησης, της διαφθοράς, το θέμα της απελευθέρωσης από το καθεστώς των θεωρήσεων. Μιλήσατε πέραν αυτών και για τις σχέσεις με τη Σερβία και για το διάλογο. Μιλήσατε με θετικό τρόπο για τις αξίες αυτές. Φυσικά, απότερο στόχος της συζήτησης αυτής είναι να αναγνωριστούν αλλήλως τα δύο κράτη. Είπατε ότι το 2013 όταν επιτεύχθη αυτή η συμφωνία για την, ε, το καθεστώς της σερβικής ε, κοινότητας στο Κωσφοπαίδιο, ε, έκτοτε δεν έχει σημειωθεί ιδιαίτερη πρόοδος. Θα πρέπει να ληφθούν λοιπόν κάποια πρωταβήματα για την αμοιβαία αναγνώριση και την πιο καλή ρύθμιση της κατάστασης. σε ό,τι αφορά το καθεστώ των συνομιλίων μεταξύ των, του Κωσυφοπαιδίου και τη Σερβία, τι γίνεται ε, για την οριστική διαθέτηση του ζητήματο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ράντο. Και τώρα να περάσουμε στον κύριο Επιτίδιο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ε, κύριε Υπουργέ, σας καλωσορίζω και εγώ στην ε, Επιτροπή μας και ευχαριστώ για την ενημέρωση. Έχω να σας κάνω δύο ερωτήσεις. Πρόσφατα, ο πρόεδρος της χώρας σας και ο πρόεδρος της Αλβανίας έκανα μια κοινή δήλωση και μίλησαν για ένωση του Κωσυφοπεδίου και της Αλβανίας. Τι νόημα έχει αυτή η ένωση. Τι προσδοκάτε να κερδίσετε αν πραγματοποιηθεί τελικά αυτή η ένωση. Και η δεύτερη ερώτησή μου είναι η εξή. Ε, η Αλβανία, όπως το γνωρίζετε άλλωστε, εκφράζει στα πλαίσια της δημιουργίας της Μεγάλης Αλβανίας επεκτατικές βλέψεις απέναντι σε όλες τις γειτονικές χώρες μεταξύ των οποίων είναι και η Ελλάδα. Με βάση αυτό το δεδομένο και αν υποθέσουμε ότι πραγματοποιείται αυτή η ένωση που ανέφερα προηγουμένως. Πεστε μου για ποιο λόγο θα πρέπει κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις η Ελλάδα να αναγνωρίσει τη χώρα σας. Ευχαριστώ. Thank you. Sandra Ευχαριστώ ε, thank you, Mr. Minister. Κύριε Υπουργέ, θα είμαι απόλυτα άμεση. Καλωσορίζομαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά οι εντάσεις στα Δυτικά Βαλκάνια μας ανησυχούν. θα ήθελα να σας ζητήσω ο λαός σας και η χώρα σας να μην υποκύψει στη ρητορική του εθνικισμού, του υπερεθνικισμού και γνωρίζω από και από τη δική μου χώρα ότι υπάρχουν ε, περιπτώσεις όπως η Ρωσία, η Τουρκία και το ριζοσπαστικό Ισλάμ που παρεμβαίνουν στην χώρα σας, προσπαθούν να επηρεάσουν τα πράγματα και θα ήθελα να μας πείτε τι ρόλο μπορεί να έχουν παίξει. Και η τελευταία μου ερώτηση θα είναι επακριβέστερη. Μετά από την επιστροφή στο κοσφοπέδιο του Ραμούς Χαραντινάη, τι νόημα έχει η συνέχιση των διαπραγματεύσεων με την Σερβία. Thank Τέλος, η Πέτερλε και Κούκαν. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για τις ξεκάθαρες απόψεις σας. Νομίζω ότι η κατάσταση είναι ε, χειρότερη από το ότι την περιγράψατε, το ότι βρίσκεται δηλαδή σε μια πραγματική αδράνεια. Νομίζω ότι τα πράγματα δεν είναι απλά στάσιμα, αλλά πηγαίνουν προς τα πίσω. Χειροτερεύουν ουσιαστικά. Πριν από 25 χρόνια είχαμε αναλάβει πάρα πολλές υποχρεώσεις και ε, δεν μπορούμε να τις φέρουμε εις πέρας. Είναι λοιπόν ευθύνη μας και καθήκον μας ε, να προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε αρνητικές εξελίξεις. Κάποιες από τις ε, ερωτήσεις μου έχουν ήδη τεθεί Θα ήθελα να θέσω όμως κάποιες ερωτήσεις τις οποίες έθεσα και στην ομάδα φίλων του Κωσυφοπεδίου. Προωθείται η ιδέα της ενιαίας αγοράς στα Δυτικά Βαλκάνια. Ποια είναι η αποψή σας γι' αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και ο κύριος Κοκάν τελευταίο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, σας καλωσορίζω και εγώ. Ανάμεσα στα άλλα ενδιαφέροντα που είπατε, αναφερθήκατε στην οριμότητα της ε, ε, κοινωνίας του κοσφοπεδίου, είπατε όμως ότι είναι και η νεότερη ηλικιακά κοινωνία στην Ευρώπη. Αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο για τη χώρα σας. Είναι βέβαια θετικό εφόσον χρησιμοποιηθεί και αντιμετωπιστεί με ευθύνη ε, και με σοβαρότητα. Εσείς είστε ακαδημαϊκός, πανεπιστημιακός και βλέπετε να υπάρχει, ε, πώς χαρακτηρίζεται τον διάλογο ανάμεσα στις βασικές πολιτικές δυνάμεις της χώρας σας. Σας ευχαριστώ συναδέλφοι για τις ερωτήσεις σας και τα σχόλιά σας. Έχουμε 15 λεπτά στη διάθεσή μας για να ακούσουμε τις απόψεις του κυρίου Υπουργού να προσθέσω κάτι σε αυτά τα οποία είπε ο Πέτερλε. Αυτή η πρόταση για την ενιαία αγορά των έξι χωρών της ε, περιφέρειας. 15 λεπτά παρακαλώ. Μέχρι 15 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ για όλες τις ερωτήσεις σας και για την ειλικρίνειά σας όσο και για τη μεγάλη σας υποστήριξη προς το ψυχοπαίδι. Θα προσπαθήσω όσο μπορώ να σας δώσω σαφείς απαντήσεις για όλα τα ζητήματα και τα θέματα που με ρωτήσατε. Η κυρία Λούνατσεκ ρώτησε τι κάνουμε για την απελευθέρωση θεωρήσεων διαβατηρίων και τι μπορεί να συμβεί στο κοινοβούλιο μας το προσεχές διάστημα ως προς την κύρωση της ε, οριοθέτησης των συνόρων με το Μαυροβούνιο. Θα ήθελα παρακαλώ να διευκρινίσω ότι αυτό το θέμα δεν είναι διακρατικό. Έχουμε εξαιρετικές σχέσεις εμείς με την Ποντγκορίτσα και είμαστε πολύ χαρούμενοι και περήφανοι που βλέπουμε ότι η χώρα αυτή κινείται προς την ένταξή της στο ΝΑΤΟ. Αυτό σημαίνει πολλά για το Κωσυφοπαίδιο, όχι μόνο για το Μαυροβούνιο. Και νομίζω ότι αυτά είναι τα πιο ευχάριστα νέα και οι καλύτερες ειδήσει από την περιφέρεια το 2017. Σε ό,τι αφορά το τελευταίο κριτήριο για την ε, άρση υποχρέωση θεώρησης διαβατήριων και τι κάνουμε εμείς ως κυβέρνηση γι' αυτό, Νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα συνεδριάσει το Κοινοβούλιο και θα επαναφέρει το νόμο αυτό για την κύρωση της συμφωνίας για την οριοθέτηση των συνόρων και ελπίζω να έχουμε αρκετές ψήφους ώστε να εξασφαλίσουμε την πλειοψηφία και να περάσει από το Κοινοβούλιο που είναι η τελευταία κρεμότητα. Ως κυβέρνηση έχουμε αυτή την πρόθεση, αλλά ειλικρινά Είμαι πάρα πολύ απογοητευμένος γιατί έχει αναβληθεί αυτό το θέμα χρόνια ολόκληρα τώρα. Αλλά εσείς τα γνωρίζετε καλύτερα από μένα. Ποια είναι η δυναμική ενός κοινοβουλίου. Και αυτά δεν πρέπει να τα σχολιάζει ένας ε, γιατί είναι διακριτή η ρόλη. Ο κύριος Αντάκτουσον ρώτησε κάτι για την καταπολέμηση της διαφθοράς και το οργανωμένο έγκλημα. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι η προτεραιότητά μας είναι και παραμένει ως κυβέρνηση το κράτος δικαίου. Και ήδη έχουμε επιτύχει πολλά. Και η Ευρωπαϊκή ε, Αποστολή EULEX μέχρι τώρα μας έχει υποστηρίξει πάρα πολύ. Αλλά ως κυβέρνηση είμαστε προσιλωμένοι ε, στην προσπάθεια αυτή και είναι βασική μας ε, προτεραιότητα. Οι εισαγγελίες, η δικαιοσύνη, η αστυνομία μας έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά τα τελευταία χρόνια, τους τελευταίους μήνες. Προχωρήσαμε ε, στη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για ένα ε, μητρό και ήρθε και η κυρία Μογκερίνη ε, στην Πρίστινα και είπε η τελευταία εκκρεμότητα, το τελευταίο θέμα προς επίλυση είναι το ζήτημα των συνόρων με το Μαυροβόνιο και μέχρι τώρα οι επιδόσεις μας και στην καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος έχουν αναγνωριστεί. Σε ό,τι αφορά την ερώτηση του κυρίου Φρόιντ για το ρόλο της Ρωσίας, αν διαδραματίζει ένα ρόλο και αν επηρεάζει τα πράγματα στο κοσυγοπαίδιο, καθόλου. Διότι το πλαίσιο μας και το πολιτικό και το πολιτιστικό στην εσωτερική μας πολιτική σκηνή είναι ε, τέτοιο που δεν προσφέρεται. Αλλά στην περιφέρεια ε, την ευρύτερη υπάρχουν χώρες που συνεργάζονται. Φέρει η Ρωσία με την Σερβία. Έχουν φτιάξει πρώτη στρατιωτική βάση στη Νίσ, που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Σερβίας και δεν απέχει πολύ από το Κωσυφοπέδιο, το Μαυροβούνιο, τη Βοσνία, τη Βουλγαρία και αυτό μας ανησυχούν. Το 2000, εκείνη την εποχή, ο πρόεδρος Πούτιν ήταν πρωθυπουργός της Ρωσικής Ομοσπονδίας και επισκέφθηκε την περιοχή συμμετέχοντας στο Ζάγκρεπ σε μία περιφερειακή σύνοδο κορυφής. Και για πρώτη φορά δημόσια δήλωσε ότι για τη Ρωσία μετά τον Ευξηνοπόντο και την περιφέρεια εκείνη, τα Βαλκάνια είναι η δεύτερη προτεραιότητά της στην εξωτερική πολιτική. Εκείνη την εποχή δεν τον λάβα πολύ σοβαρά υπόψη αυτό, αλλά την τελευταία διετία, τριετία βλέπουμε την ιστορία να επαναλαμβάνεται. Και αυτό μας ανησυχεί. Και όταν μίλησα για τρίτους παράγοντες και για γεωπτικούς ανταγωνιστές της δύση στα Βαλκάνια, τη Ρωσία είχα στο μυαλό μου. Νομίζω ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί όλες τις οδούς τις διπλωματικές, τις οικονομικές, τα ενεργειακά, ακόμα και ήπιες μεθόδους για να επηρεάσει την περιοχή. Και επειδή η περιοχή είναι ακριβώς ε, μετέωρη, ε, είναι σε μία δράνεια και κρεμότητα, αυτό ευνοεί τις δραστηριότητες της Ρωσίας και την παρουσία της στην περιοχή. Γι' αυτό το να έχουμε την δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι θέλει να φέρει κοντά της όλη την περιοχή και στο ΝΑΤΟ είναι πάρα πολύ κρίσιμο για μας. Και καμιά φορά μπορεί σε κάθε κράτος μέλος να ε, κυριαρχεί μια άλλη εσωτερική επικαιρότητα, αλλά δεν θα πρέπει να χαλαρώσετε την προσοχή σας για να σκεφτούμε πού θα βρίσκεται η περιοχή μας μετά από 10 χρόνια. Θα μπορούσα να επεκταθώ, αλλά μου είπε ο Πρόεδρος ότι δεν έχω αρκετό χρόνο και θέλω να σας απαντήσω ε, σε όλες τις ερωτήσεις. Ο κύριος Νάρτ ρώτησε για την κατάσταση στη Μακεδονία. Για το Κωσυφοπέδιο είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η χώρα. Και εμείς θέλουμε να τη δούμε να πετυχαίνει. Τι συνέβη όμως εκεί και ποιες είναι οι σχέσεις μας με την κυβέρνηση είναι πολύ καλές. Ο Νικόλα Ποπόφσκι είναι πολύ καλός μου φίλος και έχουμε πολύ καλές σχέσεις και μιλούμε και καθημερινά. Αλλά η εσωτερική κατάσταση στη Μακεδονία, όχι μόνο το τελευταίο τρίμηνο, αλλά για χρόνια τώρα, είναι μία πόλωση στο εσωτερικό της κοινωνίας. Από τη μια έχουμε τη μακεδονική κοινότητα και τη μακεδονική εσωτερική πολιτική και δεν έχει σχέση με εξωτερικούς παράγοντες, είτε είναι ε, το κοσυφοπαίδιο είτε κάποια άλλη. Έχουν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις τα δύο πολιτικά κόμματα. Και το θέμα είναι υπάρχουν αρκετοί δημοκρατικοί θεσμοί που να ε, επιτρέπουν να βρεθεί μια δημοκρατική λύση σε μια μετεκλογική περίοδο. Και δεν νομίζω ότι αυτά που συμβαίνουν τώρα και διαδραματίζονται μεταξύ των δύο πολιτικών κομμάτων δεν θα πρέπει κάποιος να προσπαθεί να τα παρουσιάσει ε, ως να ε, υπήρχε απόπειρα ε, ανάμειξη του Κωσυφοπεδίου ή της Αλβανίας στα εσωτερικά ζητήματα της Μακεδονίας. Ταυτόχρονα όμως εκεί υπάρχει μια αλβανική κοινότητα που δεν είναι μειονότητα, είναι πάνω από το 30% του πληθυσμού. Αν είναι μειονότητα, είναι μεγάλη μειονότητα και θα πρέπει να συμμετέχουν στα κοινά, στη δημόσια ζωή, σε όλα τα επίπεδα της διακυβέρνησης. Και στον 21ο αιώνα, πιστεύω, μια κοινότητα που δημογραφικά είναι το 30% ενός πληθυσμού, δεν είναι δυνατόν να μην μπορεί να χρησιμοποιεί τη γλώσσα της σε κεντρικό επίπεδο σε επίσημη γλώσσα. Αυτό είναι ένα θέμα που θα πρέπει να μας προβληματίσει και εδώ. Πάντως, εμείς ενδιαφερόμαστε πάρα πολύ να συμμετέχουν οι Αλβανοί στη Μακεδονία στην δημόσια ζωή, στην οικονομική ζωή της χώρας και η χώρα να κινηθεί προς την ένταξή της στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι δικές μας σχέσεις είναι εξαιρετικές και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τις διατηρήσουμε και να τις ενισχύσουμε. Και έχουν και πολύ καλή οικονομική συνεργασία οι δύο χώρες. Η κυρία Σουίτσα ρώτησε για τις σχέσεις Τουρκίας-Κωσυφοπεδίου. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσω απόλυτα ότι έχουμε άριστες σχέσεις με την Τουρκία. Είναι πολύ σημαντικός παράγων η Τουρκία, όχι μόνο στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, αλλά και διεθνώς. Έχουμε ανταλλαγές, οι δύο κυβερνήσεις, αλλά κατά την άποψή μου κυκλοφορεί και ένας μύθος καμιά φορά για τις τουρκικές επενδύσεις στην περιοχή μας. Αν συγκρίνετε τα στοιχεία δεν νομίζω να διαφέρουμε πάρα πολύ ή να ανησυχούμε. Ο κύριος Ράτος ρώτησε για το διάλογο. Και πώς βλέπουμε να εξελίσσεται μελλοντικά. για το διάλογο με την Ευρωπαϊκή Ένωση και για το διάλογο με τη Σερβία. Είναι ε, προς όφελός μας να εφαρμόσουμε τη συμφωνία για τη σερβική κοινότητα του Κωσυφοπεδίου και είναι και υπέρ της σερβικής κοινότητας. Και για να είμαι απολύτως ειλικρινής, δεν ανησυχούσε ποτέ το Κωσυφοπέδιο για το επίπεδο των δικαιωμάτων το οποίο θα πρέπει να χαίρουν οι Σέρβοι που ζουν στο Κωσυφοπέδιο. Σήμερα οι Σέρβοι και οι Κωσοβάροι έχουν ευρύτατα δικαιώματα. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για τα Βαλκάνια, αλλά για την Ευρώπη ολόκληρη. Ταυτόχρονα όμως θέλουμε και τους Σέρβους του Κωσυφοπεδίου να μην είναι το μακρύ χέρι της Σερβίας στο Κωσυφοπέδιο και να μην τους χρησιμοποιεί η Σερβία για να επεμβαίνει στα θέματα του Κωσυφοπεδίου. Γι' αυτό θέλουμε ε, να προωθηθεί η ένωση των ε, Δήμων και Κοινοτήτων, αλλά να υποσυρίζει τους Σέρβους του Κωσυφοπεδίου να συμμετέχουν στην κοινωνία του Κωσυφοπεδίου όμως και να μην τους διχάζει και να τους αποσπά από την υπόλοιπη κοινωνία. Νομίζω ότι έχουμε πολύ καλή πρόοδο επιτύχει. Δέκα δήμοι που είχαν Σέρβους δημάρχους ε, ε, υπάρχουν και έχουν και 10-11 έδρες στη Βουλή μας. Επειδή και οι δύο καταγόμαστε από την περιοχή αυτή, και ο κύριος Ράντος και εγώ, η Σερβία δεν είχε ποτέ τη φιλοδοξία να υποστηρίξει τους Σέρβους που ζούσαν στη χώρα, ε, να είναι τμήμα της χώρας, στην Κροατία, στη Βοσνία, ε, στο Κοσφοπέδιο, αλλά προσπαθεί να τους χρησιμοποιεί ε, ως μοχλό ανάμειξης της στα εσωτερικά όλων αυτών των χωρών. Πώς βλέπω αυτόν το διάλογο στο μέλλον. Σε ένα ορίζοντα δύο με τριών ετών θα πρέπει να συζητήσουμε με τη Σερβία και να καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία. Με στόχο την ένταξή μας στα Ηνωμένα Έθνη, με στόχο την αμοιβαία αναγνώριση των δύο κρατών και με στόχο επίσης κάποιο είδου συμφιλίωση, μια διαδικασία συμφιλίωσης. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπογράψουμε η Νευτική Συμφωνία. Αλλά το κοσμοπέδιο είναι ανεξάρτητο κράτο και ο διάλογος αυτός δεν έχει να κάνει με το καθεστώς του κοσμοπεδίου, ούτε με την κυριαρχία του. Μέχρι τώρα έχουμε επικεντρωθεί σε κάποια τεχνικά ζητήματα, έτσι, με ρεαλισμό, και θέλουμε σε ένα δεύτερο στάδιο να προχωρήσουμε και στην αμοιβαία αναγνώριση και στην ένταξη στα Ηνωμένα Έθνη. Αν δεν γίνουν όλα αυτά δεν έχει νόημα ο διάλογος και δεν έχει και χρησιμότητα, ούτε καμία ωφέλεια. Είναι ιστορική αυτή κληρονομιά, η ε, εξομάλυση των σχέσεων των δύο χωρών. Ο κ. Επιτίδιος, και ελπίζω να λέω σωστά το όνομά σας, Επιτίδιος, πριν από πάρα πολλά χρόνια είχα κάνει αρχαία ελληνικά, όταν σπούδαζα στη Βιέννη και μάλιστα μπορούσα να μεταφράσω και πλάτωνα στα γερμανικά τότε, εκείνη την εποχή. Είμαι μεγάλος θαυμαστής της χώρας σας και του πολιτισμού σας. Συμφωνώ απολύτως. Σε σχέση με τη δεύτερη ερώτησή σας, όχι την πρώτη. Η δεύτερη ερώτηση για ποιο λόγο να αναγνωρίσει η Ελλάδα το κοσυφοπαίδιο. Διότι δεν έχετε κανένα λόγο να μην αναγνωρίσετε το κοσυφοπαίδιο. Ούτε με όρους εσωτερικούς, ούτε με όρους περιφερειακούς. Νομίζω ότι το Κωσοφοπέδιο είναι μια νεοσύστατη χώρα. Ιστορικά, ανέκαθεν, είχαμε πολύ καλές σχέσεις. Και η αναγνώριση είναι μια καλή πλατφόρμα για να ενισχύσουμε τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Και είμαι πολύ περήφανος που οργανώσαμε στην Πρίστινα ένα οικονομικό φόρουμ Έλληνες επιχειρηματίες πριν από δύο μήνες και είναι τεράστιο το ενδιαφέρον των ε, Ελλήνων, της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας να έρθει να επενδύσει στο κοσυφοπαίδιο. Και έχουμε και πάρα πολύ καλές διεθνείς σχέσεις, έτσι, σε θεσμικό επίπεδο για τη Μεγάλη Αλβανία και όλο αυτό το αφήγημα, για να είμαι ειλικρινής, Αυτή δεν είναι η βασική μας ανησυχία το βασικό μας μέλημα στο Κωσυβοπαίδιο. Είμαστε χώρα ανεξάρτητη και θα παραμείνουμε ανεξάρτητο κράτος και θέλουμε να έχουμε σχέσεις και με την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ισχυρές και με όλες τις υπόλοιπες χώρες της περιοχής. Η κυρία Καλνιέτε νομίζω ρώτησε στη συνέχεια αν θα συνεχίσουμε τις συνομιλίες. Μετά την απελευθέρωση του Ράμος Χαραντινάη. Βεβαίως, ο διάλογος είναι πάρα πολύ σημαντικός και θα συνεχιστεί. Αλλά το σημαντικότερο ποιο είναι. Να υπάρχει σαφήνεια ως προς το στόχο ε, της ε, συμφωνίας και του διαλόγου. Μέχρι τώρα έχουμε επιτύχει κάποιες συμφωνίες. οι οποίες εφαρμόζονται μερικές και άλλες πάλι όχι και θα πρέπει να εστιάσουμε και στην εφαρμογή και σε ένα δεύτερο στάδιο του διαλόγου όπως σας είπα προηγουμένως. Ο κύριος Πέτερλε με ρώτησε για την κοινή αγορά. Θέλω και πάλι να είμαι απολύτως ειλικρινής. Αν υπάρχουν κάποιες χώρες στην περιοχή που έχουν συμφωνίες ελευθέρω εμπορίου με τη Ρωσία, Κάποιος προτείνει να έχει ελεύθερη αγορά. Αυτό θα είναι επέκταση της ευρωπαϊκής αγοράς ή της ρωσικής άραγε. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό γεωπολιτικό ζήτημα και ερώτημα. Το κοσυφοπαίδιο αντιτίθεται στην ιδέα αυτή. Διότι η της ρωσικης αραγε αυτο ειναι παρα πολυ σοβαρο γεωπολιτικο ζητημα και ερωτημα το κοσυφοπέδιο αντιτιθεται στην ιδεα αυτη διοτι η σερβια και η Βοσνία ακόμα δεν μας έχουν αναγνωρίσει. Και λόγω της πολιτικής μη αναγνώρισης υπάρχουν πολλά προσκόμματα για εταιρείε δικές μας επιχειρήσεις σε αυτή την περίπτωση. Η Βοσνία επέβαλε και θεώρηση διαβατηρίων τώρα για πολίτες του Κωσυφοπεδίου. Ούτε καν στο Σέγγεν δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε ελεύθερα. Και πού είναι η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, των υπηρεσιών, των κεφαλαίων και των αγαθών. Τι νόημα, αν δεν έχει όλες αυτές τις ελευθερίες, τι νόημα θα είχε μια περιφερειακή ε, αγορά. Και υπάρχει ένας φόβος στα Βαλκάνια, όχι μόνο στην Πρίστινα, ότι αυτή η κοινή αγορά είναι ένα είδος υποκατάστατου για την πολιτική διεύρυνση. Και εγώ θα σας ε, παρακαλούσα να υποστηρίξετε τις χώρες μας να κάνουν εσωτερικές μεταρρυθμίσεις. Εμείς μόλις υπογράψαμε τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και αυτό που προέχει τώρα και είναι σημαντικό να εφαρμόσουμε αυτή τη συμφωνία και να μην χάνουμε χρόνο ε, σε θέματα όπως είναι η κοινή αγορά και τέτοια. Και η τελευταία ερώτηση που έγινε από τον κύριο Κούκαν. Ήταν. Α, και η κυρία Γουόρτ, ναι, για τα θύματα, λέει ο πρόεδρο, τα, τα θύματα σεξουαλική βία. Ναι, για μα είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα και λεπτό και ευαίσθητο. Το σημειώνω αυτό που με ρωτήσατε και θα το συζητήσω με την κυβέρνησή μας. Κράτησα σημειώσει Είναι για μα σημαντική προτεραιότητα ω κυβέρνηση να υποστηρίξουμε τα θύματα πολέμου. Και υπάρχουν πολλές ομάδες που ήταν θύματα πολέμου και πολλά στρώματα. Και ο νυν πρόεδρος Θάτσι, αλλά και ο προηγούμενος πρόεδρος μας είχαν ίδιος προτεραιότητα. Και ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο κύριος Χέικ, ε, το ε, είχε κινήσει και το Ηνωμένο Βασίλειο διαδραματίζει ένα ρόλο διεθνώς. Είναι πολύ σημαντικό πάντα να τα βλέπουμε αυτά τα ζητήματα. Ζητώ συγγνώμη που ξέχασα να απαντήσω στην ερώτηση αυτή. Η τελευταία λοιπόν ερώτηση ήταν του κυρίου Έντουαρτ Κούκαν, ο οποίος είναι μέγας υποστηρικτής του Κοσφοπεδίου, αλλά και των Βαλκανίων γενικότερα. Είναι γεγονός ότι το, το έχει την πιο ζωηρή, ζωντανή και ανθούσα κοινωνία. Όχι μόνο λόγω δημογραφίας, αλλά και λόγω του εσωτερικού μας πλαισίου. Δηλαδή, από τον Ιούνιο του 1999 μέχρι το 2007-2008 αλλά και μετά στο Κωσυφοπαίδιο υπήρχε μια μεγάλη παρουσία της διεθνούς κοινότητας και αυτό ήταν πρωτόγνωρο για μας. Εξού και αυτός ο σύγχρονος και ζωντανός χαρακτήρας. Και το δεύτερο στοιχείο είναι ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλη διασπορά Κωσοβάροι ζουν από την Νορβηγία μέχρι την Νότια Αφρική και από την Πορτογαλία μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ακριβώς εξ αυτού του λόγου η κοινωνία μας πιστεύω δεν είναι η κοινωνία που είχαμε πριν από 20 χρόνια. Και προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε αυτό το κοινωνικό κεφάλαιο όχι απλώς για να βελτιώσουμε την οικονομική μας κατάσταση αλλά και για να ενισχύσουμε την ε, πολιτική κουλτούρα, τον πολιτικό πολιτισμό στο Κωσυφοπαίδιο. Πώς συνεργάζονται τα πολιτικά κόμματα, πώς συζητούν για μεγάλα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Όπως γνωρίζετε, πολύ συχνά η εξωτερική πολιτική χρησιμοποιείται ως πλατφόρμα για εσωτερική κατανάλωση, για εσωτερικούς σκοπούς. Ως κοινωνία όμως εμείς ακόμα παραμένουμε συνεκτικοί και έχουμε και μεγάλες ελπίδες. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι. Και γι' αυτό θα επιτύχει το κοσφοπέδιο. Δεν θα πω από εδώ στην αντιπολίτευσή μας τι πρέπει να κάνει. Όταν είμαστε στη Βουλή μας έχουμε δημοκρατικές ε, ε, συζητήσεις και ανταλλαγές απόψε. Ευχαριστώ στα αλβανικά. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ, Υπουργέ, και εκτιμούμε ιδιαίτερα την ε, ειλικρινιά σας στη σημερινή συζήτηση. Ελπίζουμε μετά. να έχουμε και μελλοντικέ τέτοιε ανταλλαγέ απόψεων μαζί σα. Θεωρώ ότι ήταν πολύ χρήσιμη και ωφέλιμη αυτή η ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών. Σα ευχόμαστε καλή τύχη. Ε, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα τελευταία βήματα προ την απελευθέρωση από το καθεστώ του θεωρήσεων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. Right, to... Κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στο 18 ο της ημερησίας διάταξης, μια ενημέρωση για την επίσκεψη της Επιτροπής ΑΦΕΤ στο Πακιστάν. Νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε και πολύ σύντομοι. Η επίσκεψη της Επιτροπής ΑΦΕΤ στο Πακιστάν από 18 έως 21 Απριλίου 2017 συμπεριέλαβε 8 μέλη της Επιτροπής μας, ε, η υπέροχη 8. Και οι 8 ήταν υπέροχοι. Uh, Bashir, Jean Lambert and me και υποφαινόμενο. Η αποστολή μα λοιπόν είχε πάρα πολύ έντονο πρόγραμμα και πυκνό πρόγραμμα στο Ισλαμαμπάντ και αλλού και επισκεφθήκαμε πάρα πολλού ε, αξιωματούχου του ε, Κοινοβουλίου ε, του Πακιστάν αλλά και εκπροσώπου τη κοινωνία των πολιτών και Think Tanks. Θα, βρείτε και στο, στη σελίδα του τη ΑΦΕΤΕ μια σχετική αναφορά με το Ισλαμαμπάτ. Συναντηθήκαμε με ειδικό σύμβουλο του Πρωθυπουργού για θέματα εξωτερικών υποθέσεων, με τον κύριο Κουραντούς Σκραντσκάν, ε, επικεφαλής του Εμπορικού Επιμελητηρίου και του, τον κύριο Γεσοντίκ, ε, πρόεδρο τη συμβουλή, ε, ομολόγου από τι αντίστοιχε πέντε επιτροπές της Βουλής που για πρώτη φορά συναντήθηκαν σε κοινή σύνθεση Επίσης με τον αξιωματικό Τσαντζούα, ο οποίος είναι Εθνικός Σύμβουλος Ασφαλείας και τους ηγέτες των τριών βασικών ε, κόμματων της αντιπολίτευσης του ΕΛΚ, του Πακιστανικού Κινήματος Δικαιοσύνης και τον κύριο Φαρουξαντά από την, το κίνημα MQM και με άλλους ε, συνομιλητές στην Πέσοβα επισκεφθήκαμε ένα κέντρο επαναπατρισμού για Αφγανούς πρόσφυγες του ΟΗΕ και άλλες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνδεθήκαμε με τον επικεφαλής ε, της τοπικής βουλής ε, και τέλος τελευταία ημέρα η αποστολή συναντήθηκε με τον κύριο Λόγουα Μπαλκάμα ε, της Περιφερειακής Βουλής και τον κύριο και τον κύριο εκπρόσωπο της κυβέρνησης της, ε, του Κοινοβουλίου της Πούντζαπ και ε, πρέπει να σας πούμε σε ό,τι αφορά τα θέματα πολιτικής αναφερθήκαμε στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Πακιστάν και του νέου κέντρου και πλάνου μάλλον σχεδίου πολιτικής που καταστρώθηκε φέτος. Αναφερθήκαμε σε κοινά συμφέροντα, κοινέ προκλήσεις όπως είναι οι οικονομικές σχέσεις, η κατάσταση ασφαλείας, το θέμα του κράτους δικαίου, της καλής διακυβέρνησης, σχέση ε, μεταξύ πολιτικού και ασιατικού σκέλους, ε, σχέσεις με την Ινδία, το Αφγανιστάν και την Κίνα, αλλά και με τις ΣΥΠΑ και τις χώρες του Περσικού κόλπου και θέματα ε, ασφάλειας, όπως η καταπολέμηση της ε, και η ασφάλεια στην περιοχή. Ήταν πολύ καλή η αποστολή πολύ καλή διοργάνωση και θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε για την ε, φιλοξενία του στου Πακιστανου ομολόγου μα. Αυτά από πλευρά τη ενημέρωση για την επίσκεψη τη Επιτροπή ΑΦΑΤ στο Πακιστάν. Θέλει κανεί να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Παρουσιάσατε με σωστό τρόπο τις δραστηριότητές μας Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η επίσκεψη αυτή. Θέλω να ευχαριστήσω τη Γραμματεία και τις ομάδες μας στο Μπάντα. σε ένα περίπλοκο πλαίσιο. Η συγκυρία ακολουθούσε την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για τα έγγραφα τα λεγόμενα Panama Papers Νομίζω ότι οι επαφές που είχαμε με την κυβέρνηση ήταν ουσιαστικές, ποιοτικέ. Οι μετακινήσεις δεν ήταν εύκολες, αλλά νομίζω ότι φώτισαν με ενδιαφέροντα τρόπο την κατάσταση εκεί και στην Πεσαβάρ και στη Λαχώρη. Κατανοήσαμε την περιπλοκότητα του Πακιστάν και την περιπλοκότητα της χώρας αυτής γενικά. Από πλευράς μου, στα πλαίσια αν θέλετε αυτής της αποστολής αυτό που θα ήθελα να πω όντας μέλος και της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Υποεπιτροπής Ασφαλείας νομίζω ότι θα πρέπει να εμβαθύνουμε το θέμα της προβληματικής της ασφάλειας νομίζω ότι πολύ σωστά οι ευρωπαϊκές αρχές στο Πακιστάν δεν θέλησαν να χαθούμε λίγο σε θέματα περίπλοκα, γιατί υπάρχουν και άλλα θέματα, όχι μόνο η ασφάλεια, αλλά το θέμα της ασφάλειας είναι κάτι το οποίο θα έλεγα πρέπει να μας απασχολήσει. Το θέμα ας πούμε των πυρηνικών όπλων, το θέμα της περιφερειακής συνεργασίας με τις γειτονικές χώρες, είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει επίσης να μας απασχολήσει. Θα πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή να υπάρξει μια αποστολή η οποία να έχει επαφές και με τους στρατιωτικούς στο Πακιστάν. Δεν είναι εύκολο αυτό, αλλά είναι χρήσιμο θα έλεγα για να ολοκληρώσουμε την προσπάθεια που κάναμε. Ευχαριστώ για μια ακόμη φορά τους οργανωτές. Ευχαριστώ τον κύριο Ντανζόν που δεν πέρασε τα δύο λεπτά. Ο κύριος Μαμίκης έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε και δεν θέλω να επαναλάβω τα όσα είπατε και εσείς και ο κύριος Ντανζό. Εγώ θα ήθελα να επικεντρωθώ σε τρία σημαντικά θέματα. Καταρχάς, είναι πάρα πολύ θετικό το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει την εκπαίδευση στο Πακιστάν. κατασκευάσαμε ένα σχολείο για κορίτσια ε, θηλαίων στην Πέσοβα. Και ήταν πραγματικά πάρα πολύ ενθαρρυντικό το ότι διαπιστώσαμε ποια ήταν η επιθυμία τους για σπουδές. Και είναι σημαντικό να ε, υποστηρίζονται αυτά τα σχόλια για κορίτσια, γιατί είναι στο στόχο των επιθέσεων καθημερινά, αλλά καθημερινά επιτελούν το έργο τους. Κάτι άλλο στο οποίο θα ήθελα να επικεντρωθώ. Οι συνάδελφοί μα, οι Πακιστανοί, τονίζουν τη σημασία μιας συμφωνία ε, ελεύθερου εμπορίου στην Επιτροπή ΑΦΕΤ και στην Επιτροπή Εμπορίου. Θα πρέπει να τα συζητήσουμε αυτό και να το προωθήσουμε ως αίτημα. Τρίτον, το θέμα των προσφύγων ασφαλώς. 10 χιλιόμετρα από την Οσόα επισκεφθήκαμε ένα στρατόπεδο προσφυγικό και μιλήσαμε με ανθρώπους που επί 25 χρόνια είναι στο στρατόπεδο αυτό και βλέπουμε λοιπόν πως ε, υπερασπίζονται τα ζητήματα αυτά και πώς αντιμετωπίζουν το θέμα των Ταλιμπάν. Αυτό είναι τμήμα της, του θέματος της ασφαλείας, το οποίο ανέφερε ο προηγούμενος συμπελετής και νομίζω ότι θα πρέπει να ευχαριστήσουμε όλους όσοι, όσοι διοργάνωσαν την αποστολή αυτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Μαμίκινς, λέει ο πρόεδρος, και τώρα ο κύριος Πασίρη έχει το λόγο. Παρά το γεγονός ότι αναγκάστηκα να επιστρέψω μετά την πρώτη μέρα της αποστολής, πρέπει να πω ότι ήταν πάρα πολύ καλή η αποστολή, πάρα πολύ καλά διοργανωμένη και συναντηθήκαμε με κάποιους από τους βασικούς πολιτικούς ευθύνοντες, εκτός από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος ε, έκανε πίσω την ε, ημέρα της συνάντησης, ε, γιατί υπήρξε αυτή η πολύ σημαντική δικαστική απόφαση που έλεγε εκείνη την ημέρα. Αλλά μιλήσαμε με τους πρόεδρους της Βουλής, με τον εμπορικό γραμματέα, και άλλους ομολόγους και η προθυμία των βασικών πολιτικών ηθινόντων να παραβρεθούν και ο ανοιχτός χαρακτήρα με τον οποίο ήταν μεταθυμένοι να μιλήσουν για όλα τα θέματα που μας απασχόλησαν ήταν πραγματικά πολύ ενθαρρυντικός γιατί τίποτα δεν το παρέλειψαν, τίποτα δεν το άφησαν κατά μέρος και δεν προσπάθησαν να το αποφύγουν και αυτό πραγματικά είναι εξωσημείωτο και θα πρέπει να συνεργαστούμε προκειμένου να είναι πιο εντελεχής και ευρία αν θέλετε, συνεργασία μεταξύ Πακιστάν και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι η στρατηγική εμπορική σχέση την οποία επιδιώκουν και προς την οποία κινούμαστε ή πρέπει να κινηθούμε, εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι θα πρέπει να αποστείλουμε και πρόσκληση προς τον Πρωθυπουργό της χώρας να μας επισκεφθεί. Γιατί όποτε έχουν έλθει εδώ οι ηγέτες διαφορών χωρών, αυτό έχει οδηγήσει σε μεγαλύτερη κατανόηση και, αν θέλετε, ε, παραμερισμό και οποιοδήποτε διαφωνιών και συγχύσεων επικρατούν. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάρα πολύ χρήσιμη αυτή η επίσκεψη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να περάσουμε και στους τελευταίους τρεις συναδέλφους Ράντος, Λάμπερτ και η κυρία Γκίλ. Και ο κύριος Και ο πολλανός συνάδελφος ο κύριος Γιουρέκ. Πολύ ωραία. Αυτά. Μετά όμως κλείνει ο κατάλογος. Πέντε συνάδελφοι. Ο κύριος Ραντός. ima oko 200 milijuna stanovnika. Κοιτάξτε. Α, οκ. Okay. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Ε, Νομίζω ότι με πάρα πολύ καλό τρόπο την επίσκεψή μα. Το Πακιστάν αποτελεί μια πάρα πολύ σημαντική χώρα με πάρα πολλές εσωτερικέ δυσκολίε και προκλήσει. Η τελευταία αλλαγή ισχύω ήταν δημοκρατική στη χώρα και ελπίζουμε αυτό να συμβαίνει και πάντα στο μέλλον. Η χώρα είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά αντιμετωπίζει και σημαντικά ζητήματα με την Ινδία, με το Κασμίρ και επίσης είναι γειτονική χώρα του Αφγανιστάν, το, το οποίο αποτελεί ε, α, χώρα καθόλου σταθερή. Να τονίσω κάτι που αφορά την απαγόρευση της βλασφημίας. Όταν ήμασταν λοιπόν στο Πακιστάν, τρεις γυναίκες μπήκαν στο σπίτι ενό άντρα, τον κατηγόρησαν για βλασφημία. Αυτό μάλλον πριν από 12 χρόνια έλαβε χώρα. Και τον σκότωσαν, τον δολοφόνησαν. Η εξουσία, τα πολιτικά κόμματα είναι πάρα πολύ μετριοπαθή όταν αντιμετωπίζουν τέτοια ζητήματα. Εμείς ε, το υπογραμμίσαμε το ζήτημα αυτό, αλλά πολύ φοβάμαι ότι οι σχέσεις μεταξύ στο ιστορικό της χώρας με το ζήτημα αυτό δεν είναι σαφώς ορισμένη. Και έτσι υπάρχει μεγάλη ριζοσπαστικοποίηση, η οποία μπορεί να πλήξει ιδιαίτερα στους νέους. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τώρα να περάσω στην Τζιν Λάμπερτ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, είμαι πρόεδρος της ε, αποστολής ε, της αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου με τις χώρες της Ανατολικής Ασίας. Να θέσω λοιπόν δύο-τρία θέματα. Το θέω σε ό,τι αφορά την συμφωνία GSP ε, που υπάρχει με το Πακιστάν από το 2014, όπου και υιοθετήθηκε ένας μηχανισμός από πλευρά του. σε κυβερνητικό επίπεδο και σε περιφερειακό επίπεδο για να προσπαθήσουν να προωθήσουν τις 27 σχετικές συμβάσεις. Αυτό το ακούσαμε και από τα τοπικά κοινοβούλια του, του και η Επιτροπή Ανεξάρτητων Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μας δήλωσε ότι πιστεύει ότι είναι πραγματικά χρήσιμος ο μηχανισμός αυτός και θεωρούν ότι υπάρχει πρόοδος σε θέματα νομοθεσίας, για παράδειγμα, για τα δικαιώματα των γυναικών, της βίας των γυναικών και θέματα που αφορούν τα παιδιά και άλλους τομείς. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι κάτι το οποίο προφανώς θα πρέπει να το παρακολουθήσουμε πιο ενδελεχώς μέχρι τέλους. Είναι ενδιαφέρον όμως ότι ακούσαμε κάποια σχόλια σε σχέση και με το πώς χειρίζονται άλλες χώρες το GSP+. Κάποια άλλα ζητήματα τώρα, τα οποία συζητήθηκαν. Ο διάδρομος Κίνας-Πακιστάν και ο αντίκτυπος που συνεπάγεται αυτό περιφερειακά αλλά και για τη χώρα και για τις επενδύσεις που γίνονται προς την κατεύθυνση αυτή. Περνάει με του Μπαλουτσιστάν εν μέρη και να πω ότι αυτοί που ενδιαφέρονται ιδιαίτερως έχουμε σήμερα την αντιπροσωπεία του Μπαλουτσιστάν εδώ στο Κοινοβούλιο με τους οποίους θα συναντηθούμε σήμερα το απόγευμα αν ενδιαφέρεται κανείς. Και αυτά ήταν λοιπόν σημαντικά ζητήματα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα της βλασφημίας. Αυτό το διαπιστώσαμε και λίγο πριν καταφτάσουμε. Ήταν ιστορική απόφαση στο Κοινοβούλιο. Έτσι χαρακτηρίστηκε η αναγνώριση δηλαδή της ανάγκης να αλλάξει κάπως ε, η νομοθεσία. Όχι να καταργηθεί φυσικά το μάρτυμα αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν μια αρχή. Θα πρέπει να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις προς την κατεύθυνση αυτή, εφόσον φυσικά υπάρξουν εξελίξεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, αλλά και η Πρόεδρος είναι η Ναγκίλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι θα συμφωνήσω με τους συναδέλφους Πράγματι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση που έγινε. Ήμασταν τυχεροί που πήραμε μέρος. Είναι σαφής η βούληση των Πακιστανών να εμπλακούν σε διάλογο. Οι συζητήσεις οι οποίες ήταν οι πιο καρποφόρες ήταν αυτές με την κοινωνία των πολιτών. Και νομίζω ότι συναντήσαμε αρκετούς εκπροσώπους της θα πρέπει εδώ να υπενθυμίσουμε τις ανησυχίες που εξέφρασαν για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ελευθερία έκφρασης. Όπως είπε και ο συνάδελφος για τους νόμους για την βλασφημία, ε, δύο μέρες πριν φτάσουμε λιντσαρίστηκε ένας φοιτητής γιατί κατηγορήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα. Ε, επίσης και μια καθηγήτρια εδάρια Νηλεός ε, για τον ίδιο λόγο. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το κλίμα έλλειψης ανοχής απέναντι στις θρησκευτικέ μειονότητες. Το σύστημα της δικαιοσύνης δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει, γι' αυτό πρέπει η κυβέρνηση να αλλάξει γραμμή εδώ. Οι νόμοι αυτοί για τη βλασφημία εφαρμόζονται ε, με ε, τρόπο ο οποίος είναι πολύ ευρύς και δεν προστατεύεται η ελευθερία του λόγου. Τώρα σχετικά με το GSP+. Θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε σαν μέσο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά. Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να δούμε τι δράση μπορούμε να αναλάβουμε και να προσέξουμε επίσης τι γίνεται με την χρηματοδότηση από τις χώρες του κόλπου, όπως επίσης και για την διδασκαλία του μίσους στα θρησκευτικά σχολεία, τα μέντρεσε. Κοιτάξτε, όλο και περισσότεροι συνάδελφοι παίρνουν το λόγο. Ε, έχουμε καθυστερήσει 15 λεπτά, έχουμε άλλη μία συζήτηση και έχουμε επίσης και ένα workshop που ξεκινάει στις 12.30. Εν πάση περιπτώσει, ο επόμενος είναι ο κύριος Γιούρεκ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ σύντομα να ζητήσω να μάθουμε αν έχουν υπάρξει πληροφορίες στην περίπτωση nasze relacje Να δούμε αν πράγματι γνωρίζουν ότι οι αμοιβέ σχέσει με την χώρα αυτή επηρεάζουν άμεσα την εικόνα του Ισλάμ. Το Πακιστάν πάντα θεωρεί το στην Δύση σαν πλουραλιστική κοινωνία. Και πράγματι κάποιοι νόμοι αυταρχικοί κάτω από, από το Μουσάραφ ε, και από την κυβέρνηση Μπούτο έθεσαν σε αμφισβήτηση τον πλουραλισμό αυτό. Βλέπουμε ότι τώρα υπάρχουν αντιδράσεις από πλευράς ε, ε, των μουσουλμανικών κοινοτήτων. και θα πρέπει να διασφαλιστεί ο σεβασμός της κοινωνίας των πολιτών σε όλες τις εκφράσεις. οι ευθύνες τις οποίες έχουν ε, ε, οι τοπικές κοινότητες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Mr. Κύριε Γιουρέκ, να προτείνω. Κύριε Γιουρέκ, με ακούτε. Θα προτείνω να κάνουμε μια ε, συζήτηση κατηδίαν για το θέμα αυτό αργότερα. Γιατί δεν νομίζω ότι αυτό α, θα πρέπει να αναφερθεί σε δημόσια συζήτηση της Επιτροπής ΑΦΕΤ. Είναι θέμα ίσως ε, σιωπηρή ε, διπλωματίας, αλλά παρακαλώ να επικοινωνήσετε μαζί μου, αν θέλετε, για το θέμα αυτό σε ό,τι αφορά το Πακιστάν. Και τώρα η κυρία Ζαύκο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόεδρε, νομίζω ότι τα συνοψίσατε πάρα πολύ καλά τα πράγματα στην ε, ενημέρωσή σας. Να τονίσω ένα θέμα το θέμα των 60 εκατομμυρίων γυναικών που δεν είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, δεν έχουν ταυτότητες. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πιστεύω θα πρέπει να το παρακολουθήσουμε. Επίσης θα ήθελα να συμφωνήσω με τους συναδέλφους που μίλησαν για τα ζητήματα των προσφύγων. Όταν αυτοί οι πρόσφυγες επαναπατρίζονται μετά από 30 χρόνια, κάποια από τα κορίτσια αυτά Μίλησα μαζί Δεν ε, τους επιτρέπουν να πάνε στο σχολείο και έχουν και θέματα ασφάλειας να αντιμετωπίσουν. Αυτά θα πρέπει λοιπόν να τα συζητήσουμε περαιτέρω, θεωρώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Νάτο. Θα ήθελα να ε, αφοσιωθώ στην κοινωνική κατάσταση στο Πακιστάν. Έχει ε, μεγάλη επιρροή το δόγμα Χανάφη το Μπάντι που είναι ε, ακριβώς ε, το υπόβαθρο των ε, ακραίων Ταλιμπάν. Οι περισσότεροι μετρεσέδες στα σχολεία εκεί, τα θρησκευτικά στο Πακιστάν, χειραγωγούνται από το Inter-Service Intelligence, που είναι βασικά η μυστική υπηρεσία του στρατού στο Πακιστάν. Αλλά όλα αυτά προέρχονται από μια βαθιά και πολύ σκληρή ε, ριζοσπαστικοποίηση που ε, προέρχεται ε, από αυτά τα θρησκευτικά σχολεία από όπου προέρχονται οι Ταλιμπάν και ο ακραίος Ισλαμισμός. Λαμβάνουμε υπόψη ότι το πρώτο θύμα είναι ο ίδιος ο πακιστανικός λαός. Αλλά το κοινωνικό φαινόμενο αυτό με ενισχύει πολύ περισσότερο, πολύ πιο πολύ από την οικογένεια Μπούτο, το επικοδόμημα, το πολιτικό και τα υπόλοιπα που ανήκουν στην ιστορία της χώρας. Σα ευχαριστώ και τέλος ο κύριος Γκάλερ έχει το λόγο. Σα ευχαριστώ και θα είμαι σύντομο και πολύ λυπάμαι που δεν συμμετείχα στην αποστολή. Μία ερώτηση έχω να κάνω για το σχόλιο της κυρίας ε, Νίνα Γκίλη. Αναφέρθηκε στην κυρία στην γυναίκα αυτή την Αχμάντη με την οποία συναντήθηκε. Το ερώτημα είναι κατά πόσον η Αχμάντη ήταν η μοναδική μειονότητα η οποία α, διατηρήθηκε σε διαφορετικό ε, κατάλογο ψηφοφόρων και το έχω επικρίνει αυτό στο παρελθόν. Και πέρσι ήδη άκουσα από έναν υπουργό ότι αυτός ο ε, ε, ξεχωριστός κατάλογος ψηφοφόρων για τους Αγμάντι είχε καταργηθεί. Αυτό σας το επιβεβαίωσαν στη συζήτησή σας με την εκλογική επιτροπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση αυτή, λέει ο πρόεδρος. Κοιτώ προς την ομίγυρη. Δεν νομίζω να μας ενημέρωσαν για το θέμα αυτό σε καμία περίσταση. Συμφωνείτε, συμφωνείτε. Ναι, κυρία Γκίλ, ναι, το θίξαμε το θέμα αυτό και πολλά από τις, πολλές από τις συστάσεις σας τις ε, προωθήσαμε στον επικεφαλής της ε, Επιτροπής ε, των Εκλογών. Δεν είχε εφαρμοστεί αυτό στο καταστατικό, αλλά κάποιες από τις συστάσεις σας είχαν συμπεριληφθεί και μας διαβεβαίωσαν ότι επρόκειτο να εφαρμοστούν όλα αυτά μέχρι τις επόμενες εκλογές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, συνάδελφοι, και να σας ενημερώσω ότι το έργο του Μιχαήλ Γκάλερ σε διάφορες περιστάσεις το τόνισαν και μας ευχαριστήσαν γι' αυτό. Σε διάφορες περιστάσεις, διάφοροι ομολογοί μας. Σας ευχαριστώ. Άλλα σχόλια, όχι. Να περάσουμε στο 19 λοιπόν τη ημερήσια διαταξή τώρα για τι πολιτικέ σχέσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση με την Λατινική Αμερική. Πρώτη εξετασή σχεδίου έκθεση ίδια πρωτοβουλία για τι πολιτικέ σχέσει τη Ένωση μα και τη Λατινική Αμερική και τη Καραϊβική. Ο Στόλφος Χαβιλοπές από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες είναι ο εισηγητής και χωρίς καθυστέρηση θα του δώσουν το λόγο. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω μόνο συνάδελφοι ότι θα διοργανωθεί ένα σεμινάριο για τη Μέση Ανατολή εδώ στις 12.30. Αλλά έχουμε και καθυστέρηση 40-45 λεπτά για το θέμα αυτό και τώρα το λόγο λοιπόν το δίνω παρά στον κύριο Λόπες. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε που μου δίνει το λόγο. Σύντονη παρουσίαση. Γιατί εκπονούμε αυτή την έκθεση και με ποια κριτήρια. Πώς ορίσαμε το περιεχόμενο και ποιος είναι ο πότερος στόχος, έτσι. Πρώτον, η έκθεση κατατίθεται για να δοθεί μια όθηση στη σχέση μας, γιατί η τελευταία αντίστοιχη έκθεση έγινε προεξαετίας. Ήταν η έκθεση Σαλαφράνκα που εγκρίθηκε εδώ στο Κοινοβούλιο. Αλλά τα τελευταία 6 χρόνια έχουν, συνέβη πάρα, έχουν συμβεί πάρα πολλά και στη Λατινική Αμερική και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βαθιές αλλαγές, κάποιες κρίσεις που συσσωρεύονται. Για παράδειγμα το 2010 δεν είχαμε την υπηρεσία εξωτερικής δράσης, ήταν στα Σπάργανα έχουν γίνει αλλαγές και εδώ και εκεί και τώρα μετά το Brexit είναι βαθιές οι αλλαγές αυτές. Αντίστοιχα στη Λατινική Αμερική ο κύκλος της οικονομικής αύξησης ε, ε, ε, με τη μεγέθυνση και την άνθηση των εμπορευμάτων. Έχουμε πολιτικές αλλαγές βαθιές σε κάποιες περιοχές που αφορούν και τη σχέση μας. Άρα λοιπόν τα τελευταία έξι χρόνια είχαμε πολλές αλλαγές, ε, αλλά είμαστε κοινότητα συμφερόντων, έχουμε κοινέ αξίες και μετά τις διεθνείς ε, αλλαγές που έγιναν πέρσι χρειάζεται κάποια ανανέωση λοιπόν στη σχέση μας. Η έκθεση αυτή αποκτά και ιδιαίτερη σημασία μετά την νέα κυβέρνηση των Ηνωμένων μετά το νέο διεθνές πανόραμα, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση αναζητεί εταίρους στον κόσμο που να έχουν την ίδια θεώρηση ε, για τις διεθνείς σχέσεις, για την πολυμερή συνεργασία, για τις ανοιχτές κοινωνίες, για τους κανόνες και το διάλογο ως τρόπο ευθέτησης της εξωτερικής πολιτικής. Και όχι μόνο αυτό, έχουμε και κοινό θεματολόγιο με τη Λατινική Αμερική. Εκεί εστιάζει η έκθεση, θέλει να είναι οριζόντια και επικοδομητική, πάρα πολύ σημαντικό αυτό για μας προσπαθεί να εκπέμψει το μήνυμα ότι για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στρατηγική προτεραιότητα η σχέση μας με την Λατινική Αμερική. Αυτό είναι το light motif όλης της έκθεσης. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν και συγκεκριμένες προτάσεις. Πρώτον, θα ήθελα να εξηγήσω ότι Έχουμε τέσσερις συμφωνίες επιτάπητος, πολύ σημαντικές. Πολιτικός διάλογος με την Κούβα, που ε, ξέρουμε ότι έχει πολιτικό αντίκτυπο εκεί. Διαπραγματεύσεις με τη Μερκοσούρ, τεράστια οικονομική συνεργασία. Ανανέωση των εμπορικών συμφωνιών με Μεξικό και Χιλή. Δεν είναι μόνο τα θεσμικά αυτά και οι συμφωνίες, αλλά και το κοινό περιεχόμενο που μας ενώνει και θέλουμε να μοιραστούμε. Δεν έχουμε απλώς την ίδια αντίληψη για τις διεθνείς σχέσεις, αλλά έχουμε και κοινά θέματα, κοινή ατζέντα. Μία ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, ε, δηλαδή με αναδιανομή του πλούτου, ε, καταπολέμηση των φορολογικών παραδείσων, ισότητα φύλων, καταπολέμηση των παραβιάσεων των ε, πιο ευαλώτων ομάδων. Θέματα ασφαλείας που είναι διαφορετικά ε, σε κάθε περίπτωση. Εμείς εδώ έχουμε τη δρομοκρατία, στη Λατινική Αμερική το λαθρεμπόριο ναρκωτικών. Βέβαια μπορεί να είναι διαφορετικά στις καταστάσεις, αλλά τα θέματα κοινά. Επίσης, τονίζουμε ότι η σημερινή μας ε, σχέση είναι πάρα πολύ θεσμική. έχουμε πολύ ε, ε, ε, υψηλέ σχέσει σε υψηλό επίπεδο, δηλαδή με συνόδους κορυφής, ε, την και Eurolat κτλ. Αυτό όλα τα λέμε στην έκθεσή μας και γνωμοδοτεί η Επιτροπή Ανάπτυξης. ΔΕΒΕ. Αναφέρονται και κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις, η ενευτική διαδικασία στην Κολομβία, η περίπτωση της Κούβας, αν και η βασική εστίαση είναι περιφερειακή. Γίνεται Εκεί η συζήτηση αυτή είναι η βάση της πρώτης πρότασης. Και ολοκληρώνοντας θέλω να πω ότι μια τέτοια έκθεση έχει νόημα όταν συμπίπτει η έγκρισή της με το επόμενο ε, φθινόπορο που είναι πάρα πολύ επίκαιρη ε, στη σχέση μας. Έχουμε συνάντηση κορυφής ε, στο Σαλβαδόρ αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Η Eurolat επίσης συνεδριάζει κοινοβουλευτικά και προετοιμάζεται μια νέα στρατηγική, ε, μια νέα ανακοίνωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις σχέσεις με την ε, Λατινική Αμερική. Μέχρι και η ΟΚΕ ε, γνωμοδοτεί. Θέλουμε λοιπόν να είναι η δική μας έκθεση ένα στοιχείο που θα ενταχθεί στο συνολικό θεματολόγιο του φθινοπόρου. Τα τελευταία χρόνια ε, δεν ήταν η ε, κατάσταση πάρα πολύ εύκολη. Εγώ προσβλέπω τώρα στην αγαστή συνεργασία με τις άλλες πολιτικές ομάδες και περιμένω τις τροπολογίες. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Lopez. Ευχαριστώ κύριε Λόπες. Εφτά ακόμα ομιλητές, οκτώ ομιλητές, εννέα ομιλητές. Νομίζω ότι η Λίγκουα Φράγκα το τα επόμενα 45 λεπτά θα είναι τα ισπανικά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή για το πνεύμα το οποίο διέπει την έκθεσή του. Πράγματι πρόκειται για μια συνενετική πρόταση και θα είναι ένα καλό μέσο για να πετύχουμε κάποιες πλειοψηφίες. Αυτό εύχομαι. Είναι λοιπόν μια θετική. Νομίζω όμως και πρέπει να το πω ότι είναι βελτιώσιμο. Νομίζω ότι υπάρχουν πλευρές οι οποίες πρέπει να διορθωθούν, κάποιες άλλες πλευρές που πρέπει να βελτιωθούν και νομίζω ότι υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία κατά περίπτωση θετικά και άλλα αρνητικά. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να αγνοήσουμε σαν παράδειγμα την κατάσταση της Βενεζουέλας είναι ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει πάρα πολλές συζητήσεις. Δευτερευόντως δεν θα πρέπει να περιοριστούμε εμείς ε, στην αναγνώριση των δυνατοτήτων των τοπικών μέσων, των περιφερειακών μέσων, αλλά να ε, τονίσουμε και τα προβλήματά τους. Ε, στην περίπτωση της Μερκοσούρ, σαν παράδειγμα, υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν Μέχρι τώρα έχουν δημιουργηθεί όμως σε πολλούς τομείς προβλήματα από τη μη χρήση των δυνατοτήτων. Στα θέματα της, ε, την περίπτωση Όντεμπρεχτ. Ε, λοιπόν, υπάρχουν επίσης ε, κάποιες ψευδοδημοκρατικές διαδικασίες που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε διότι οδηγούν σε απολυταρχικές καταστάσεις όπως την Ικαραγουά. Στην Κούβα υποτίθεται ότι υπάρχει ο πολιτικός διάλογος, είναι όμως σαφές ότι έχει υπάρξει στήριξη του διαλόγου αυτού, αλλά το ψήφισμα θα πρέπει να ασχοληθεί και με θέματα επιμέρους, τα οποία αξίζουν να αντιμετωπιστούν με ανεξαρτησία και κυρίως με ευθύνη, γιατί είναι σαφές ότι το καθεστώς εκεί δεν ανταποκρίνεται στα δικά μας επίπεδα. Σε επίπεδο ε, οικονομικό θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν συγκεκριμένα θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, θα πρέπει να σταθώ σε κάποια από αυτά τηλεγραφικά. Λοιπόν, η προστασία των επενδύσεων, το κράτος δικαίου, ε, τα μέτρα τα οικονομικά που πρέπει να ληφθούν και στον τομέα των φιλολογικών έτσι ώστε να βελτιωθεί η οικονομική απόδοση των χώρων αυτών Έχουμε όμως να αντιμετωπίσουμε και το θέμα της χειροτέρευσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την τρομοκρατία και ταυτόχρονα την συνεργασία μας και σε επίπεδο βοήθειας, γιατί πολλές φορές όπως στην Κολομβία και στον Περού έχουν πρέπει να προχωρήσουν ακόμα περισσότερο σε επίπεδο συνεργασίας, διότι έχουν ε, αντιμετωπίσει, να αντιμετωπίσουν πάρα πολλά προβλήματα τα οποία δημιουργήθηκαν στο παρελθόν. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τάνο και έχει το λόγο. Δεν είχα ζητήσει το λόγο, αλλά μια και μου το δίνετε. Α, ναι, αλλά πάντα σημειώνουμε το όνομά σα, λέει ο πρόεδρο. <laughs> Πάντα το σημειώνουμε το όνομά σα ε, ε, εκ των προτέρων. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα και εγώ και η ομάδα μα ήμασταν υποστηρικτέ των καλών σχέσεων με τη Λατινική Αμερική και θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή, τον κύριο Λόπες για τη δουλειά του. Σαφώς ε, αυτό που είπε κάποιος ε, πριν από κάποια χρόνια το συνδυασμένο ΑΕΠ ε, της Λατινικής Αμερικής από κοινού είναι ίσο με το ΑΕΠ της Κίνας και αυτό και σε ό,τι αφορά και την Κουβά, τη Βενεζουέλα. Έχουμε ιστορικούς δεσμούς μέσω των δύο χωρών της Πορτογαλίας της Ισπανίας και συχνά έχω μεταβεί και εγώ στην Λατινική Αμερική και ιδιαίτερο στη Χιλή, στην Αργεντινή και στην Κολομπία Και φυσικά, καλώς ορίζω την σύσφυξη των σχέσεων με την Ήπειρο και ασφαλώς ε, έχουμε τις εταιρικέ σχέσεις ε, πρώτης γενιάς μεταξύ Χιλής, Μεξικό και Ευρωπαϊκής Ένωσης και χαίρομαι που πλέον η Μερκοσούρ ε, και η Συμφωνία Μερκοσούρ μπορεί να αναστηθεί. Είναι πάρα πολύ λυπηρό για τη χώρα μου η οποία έχει ξεκινήσει να επωφελείται από τις εμπορικές αυτές σχέσεις ε, που θα γίνει το Brexit όταν ουσιαστικά ολοκληρωθεί η συμφωνία Mercosur με την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει το Ηνωμένο Βασίλειο να επαναδιαπραγματευτεί διμερείς σχέσεις με όλες αυτές τις χώρες. Και ο πρέσβης ε, της Βενεζουέλα στο Ηνωμένο ε, Βασίλειο και διάφοροι άλλοι θα δήλωσαν ότι θα διακυβευτούν όλες αυτές οι συμφωνίες με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Όλα αυτά θα πρέπει να τα σκεφτούμε προσεκτικά στα δύο χρόνια πριν τον Brexit, αλλά εγώ προσωπικά και η ομάδα μου θα υποστηρίξουμε τις ενέδωρες σχέσεις και είναι προφανές ότι η Λατινική Αμερική έχει πολύ πιο πολλά κοινά μαζί μας από πολλές απόψεις από ότι η Κίνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Τάνοκ, ο Νομίζω ότι η πρόταση του Χαβιέ είναι θετική, αλλά υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία θα ήθελα να υπογραμμίσω. Καταρχάς, εκρηκτική κατάσταση στη Βενεζουέλα δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε. Έχουμε να κάνουμε με μια δραματική κατάσταση, η οποία στην καλύτερη περίπτωση θα οδηγήσει σε ένα ανοιχτό εμφύλιο πόλεμο και στη χειρότερη ε, σε ένα πραξικόπημα, το οποίο στρατιωτικό, το οποίο ε, θα διαπράξει προφανώς αυτός ο εκλεγμένος δικτάτορας όπως ο Χίτλερ, ο κύριος Μαδούρο. Δεύτερον, ένα γενικότερο θέμα για την περιοχή είναι το θέμα της διαφθοράς. Είναι ενδημικό πρόβλημα στη Λατινική Αμερική και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με συστηματικό τρόπο θα πρέπει να στηρίξουμε την ριζικά και σε βάθος προσπάθεια διαχωρισμού των εξουσιών για να διασφαλίσουμε τον αγώνα για καταπολέμηση της διαφθοράς για την Κούβα. Η συμφωνία ανάμεσα στην Κούβα και το Ηνωμένο Βασίλειο πραγματικά με οδηγεί σε πλήρη σύγχυση, εν πάση περιπτώσει, διότι το κοθεστός της Κούβας δεν λειτουργεί μόνο κατασταλτικά, αλλά ελέγχοντας επίσης με στρατιωτικό τρόπο στο σύνολο της οικονομίας. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να γνωρίζουμε. Ε, θα έλεγα ελέγχει πλήρως ε, το, με στρατιωτικό τρόπο την οικονομία. Οπότε στην ουσία αυτό το οποίο ζητάμε να γίνει στην Κούβα ε, είναι κάτι το οποίο συνδέεται άμεσα με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ελευθεριών. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο είναι αντιφατικό με την ηγεμονία της ε, ε, καστρικής σε εισαγωγικά μορφής ελέγχου και της ε, διαδόχου αυτής καταστάσεως που κυριαρχεί πλήρως στην Κούβα. Ευχαριστώ κύριε Σκόουσο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και τον εισηγητή για αυτό. Ε, το σχέδιο έκθεσης είναι θετική, μπορούμε να τη στηρίξουμε. Είναι περιφερειακή συνεργασία, ολοκλήρωση, δίνεται έμφαση στη σχέση μας ε, με ε, την κοινότητα της Λατινικής Αμερικής. Υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν μας αρέσουν, αλλά μπορούμε να αλλάξουμε την απόχρωση λίγο. Έχουμε πλέον περιφερειακή συνεργασία, ενώ στο παρελθόν είχαμε εμπορική συνεργασία, ιδεολογικά φορτισμένη κατά την άποψή μας, ε, που δεν ε, βοηθούν την ανάπτυξη των λαών. Επίσης αναφέρεται κάποιες χώρες ενώ κάποιες άλλες όχι. Ας πούμε, τι γίνεται με την ελευθεροτυπία. 14 δημοσιογράφοι έχουν δολοφονηθεί, 7 στο Μεξικό και μόνο. Εχθές δολοφονήθηκε στο Μορέλος ένας δημοσιογράφος και στο Μεξικό έχουμε εξαφανίσει ενώ στην Κολομβία μας ανησυχούν οι δολοφονίες αγωνιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων από παραστρατιωτικές ομάδες που θέλουν να, να βαγίσει η ειρνευτική συμφωνία. Γενικά είναι θετική έκθεση και θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε γενικώ. Κύριος Ουρτάσουν των Πρασίνων. Καλημέρα σας. Ευχαριστήσουμε ε, και εμείς από πλευρά των Πρασίνων. Είναι καλό το κείμενο. Ε, ε, δίνουμε ένα μήνυμα ότι θέλουμε να δώσουμε μια νέα όθηση στην περιφερειακή συνεργασία. Ευρώπη και Λατινική Αμερική από κοινού πρέπει να δράσουν σε διεθνές επίπεδο. Τώρα που βλέπουμε να αναδύεται μια αντιδραστική διεθνής που θέλει να καταστρέψει την πολυμερή συνεργασία. Εμείς λοιπόν θα πρέπει να διατηρήσουμε την πολυμερή συνεργασία, να δώσουμε νέα όθηση συμφωνία των Παρισίων κατά της κλιματικής αλλαγής στα Ηνωμένα Έθνη κτλ. Άρα θα πρέπει να οικοδομήσουμε ε, και να βασιστούμε σε κάποια θετικά του παρελθόντος που υπάρχουν. Το ρόλο που έχουμε παίξει στην ειρηνευτική διαδικασία στην Κολομβία, νέα συμφωνία με την Κούβα, που θα κάνει την Ευρωπαϊκή Ένωση να πρωταγωνιστήσει ξανά σε αυτή τη νέα ατζέντα, την ανανεωμένη και το θεματολόγιο που λέγατε, θα μπορέσουμε και εμείς να κάνουμε κάποιες ενδιαφέρουσες ενδεχομένως προτάσεις να δούμε μια διεθνή ατζέντα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, την καταπολέμηση της ανισότητας, γιατί έχουμε ανισχυτικά στοιχεία στη Λατινική Αμερική. Έχουμε επιστοδρόμηση, το θέμα του χρέους φυσικά. Υπάρχει μια πρόαση λατινοαμερικανική για τον ΟΗΕ, για ένα πλαίσιο αναδιάρθρωσης των χρεών των χωρών και βεβαίως το θέμα της ισότητας των φύλων που σε αυτό το τομέα η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να κάνει πάρα πολλά. Από κοινού έχουμε δύο καλά εργαλεία, δύο συμβάσεις Ισταμπούλ και ακόμα μία διεθνή. Η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης είναι στο σύμβολο της Ευρώπης. Ε, επ' αυτόν λοιπόν μπορούμε να συνεργαστούμε με πολύ καλό τρόπο. Μερικά παραδείγματα σας δίνω κύριε Σιγητά που είμαι βέβαιος ότι θα σας αρέσουν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Τρεις ομιλητές έχουμε ακόμα. Κύριε Σαλαφά. Ευχαριστήσω τον εισηγητή. Έχει δώσει μια πάρα πολύ καλή βάση για να δουλέψουμε τις σχέσεις με, ε, με τη Λατινική Αμερική. Ιδιαίτερα και στα πλαίσια της ε, σύντομης, σε λίγο καιρό, εν πάση περιπτώσει, προσεχούς συνάντησης κορυφής. Νομίζω ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία όμως θα πρέπει να συμπληρωθούν. Καταρχά σε επίπεδο στρατηγικής συνεργασίας, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η συνεργασία αυτή μέσω του συστήματος των συναντήσεων σε επίπεδο κορυφής ε, γεννά κάποιες ευκαιρίες ε, και τον ε, επόμενο Δεκέμβριο θα πρέπει να εκφράσουμε την επιθυμία μας η συμφωνία αυτή να ολοκληρωθεί και να επικυρωθεί κατά τη διάρκεια της παρούσης κοινοβουλευτικής περίοδου. Τώρα ειδικά για το Μεξικό και τη Χιλή όχι μόνο θα πρέπει να είμαστε ευτυχείς για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και νομίζω ότι υπάρχει αρκετός χρόνος έτσι ώστε να ολοκληρωθεί και η διαδικασία επικύρωσης. Τώρα για τη βοήθεια για την ανάπτυξη είναι σαφές ότι κάποιες από τις χώρες αυτές ε, ε, εποφελούνται και θα πρέπει να προσπαθήσουμε και εμείς να ζητήσουμε την αναθεώρηση του κανονισμού ε, το κάτι το οποίο είναι απαραίτητο και αναφέρομαι τώρα στην ανάγκη αναζήτησης ενός μηχανισμού σε συνεργασία με τους εκπροσώπους των χωρών αυτών έτσι ώστε να προωθήσουμε με πιο φιλόδοξο τρόπο τις διαδικασίες συνεργασίας. Θα ήθελα να θέσω μια ερώτηση. Κύριε Λόπες, τι ιδέες έχετε σε σχέση με τον χρονισμό. Νομίζω ότι η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης προσπαθεί να συγχρονιστεί με τον δικό μας χρονισμό, αλλά όπως είπε στην αρχή ο εισηγητής θα μπορούσε να γίνει μια κοινή προσπάθεια και με, τις, ε, και με τα υπόλοιπα όργανα. Ευχαριστώ. Κύριος Ασής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και θα ήθελα να πω ότι και εγώ συγχαίρω τον εισηγητή, γιατί πραγματικά η έκθεση αυτή αποτελεί μια πολύ καλή βάση, επί τη οποία θα πρέπει να εργαστούμε και περαιτέρω. Αναφέρθηκε ήδη την κρίσιμη σημασία σε να θέσουμε το θέμα τη Βενεζουέλα. Πρόκειται ασφαλώ για την πιο σοβαρή περίπτωση μη σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λατινική Αμερική στην παρούσα φάση. Και εδώ γίνεται μια απόπειρα να μπει μια δικτατορία ουσιαστικά δικτατορία σωστή. Κοιτώντας και τι συμβαίνει και τις τελευταίες ημέρες, βλέπουμε ότι οδηγούμαστε προς τη σύσταση μια βολής χωρίς καν δημοκρατική βάση και σε καμία περίπτωση αυτό δεν εκπροσωπεί τη θέληση και τη βούληση του λαού της Βενεζίας. Βλέπουμε λοιπόν ότι πολύ απλά σε μια τέτοια έκθεση θα πρέπει να αποτυπωθεί και η κατάσταση στην Βενεζουέλα. Κατά δεύτερον, συμφωνώ ε, επί των βασικών αρχών, αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε πιο στενά στην κοινωνικονομική ανάλυση της κατάστασης στην Λατινική Αμερική, η οποία είναι πολύ διαφορετική, γιατί δεν είναι όλες οι χώρες διατεθειμένες να συνεργαστούν με την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι σημαντικό να διακρίνουμε τις διαφορές αυτές και να προσπαθήσουμε να τις ξεπεράσουμε. Και επίση έχουμε και άλλα ζητήματα με κάποιε χώρε τη Λατινική Αμερική, οι οποίε ενδεχομένω να μην είναι στο βαθμό της σε ό,τι αφορά τα ιστορικά του προβλήματα, αλλά υπάρχουν προβληματικέ τάσει τι οποίε θα πρέπει να τι δείξουμε. Και το θέμα τη διαφθορά, θα πρέπει να το δείξουμε, γιατί αφορά μεγάλο τμήμα τη ε, Λατινική Αμερική. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό και η Ευρώπη θα πρέπει να υποστηρίξει αυτούς που καταπολεμούν την ε, διαφθορά. Σε ό,τι αφορά την στρατηγική συνεργασία τώρα, Όπω αναφέρθηκε και από τον συνάδελφο Σαλαφράγκα, πολλά ακόμα θα πρέπει να κάνουμε. εξετάζοντα την έκθεση που προετοίμασε ο κύριο Σαλαφράγκα και που έχει καταρτήσει και σε διάφορε περιστάσει στο παρελθόν. Θα πρέπει να διαπιστώσουμε ότι πραγματικά είναι πάρα πολλά αυτά που θα πρέπει να γίνουν για να υπάρξει πραγματικά σωστή αντιμετώπιση των εκθέσεων. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο πρόεδρο, τελευταίο αλλά και τυχερό ο κύριο Μιλανμόν. Ε, Ευχαριστώ τον εισηγητή και εγώ ε, για το έργο του. Νομίζω υπάρχει συναντήληψη εδώ ευρύτατη και η έκθεση είναι θετική. Αλλά έχω και κάποια αλλά συγκεκριμένα. Τα είπαν και ο Λουίς Δεγκράντες και ο Νάτσο Σαλαφράνκα. Διαβάζοντας την έκθεση ιδιαίτερα την αιτιολογική σκέψη α και την πρώτη και δεύτερη παράγραφο βλέπω μια συγκυριακή προσέγγιση ε, στη σχέση μας και σε σχέση με τις παγκόσμιες προκλήσεις. Υπάρχει κάτι που έχουμε ξεχάσει. Έχουμε πολύ στενές σχέσεις κάθε είδους, ιστορικές, πολιτιστικές, ε, όλα τα υπόλοιπα που λέτε μπορούν να αφορούν και οποιαδήποτε άλλη περιοχή του κόσμου αλλά εμείς έχουμε πάρα πολύ πυκνές σχέσεις με τη Λατινική Αμερική. Είμαστε φυσικοί σύμμαχοι, αλλά υπάρχει και μια ιδιαιτερότητα στις σχέσεις Λατινικής Αμερικής με πολλές ευρωπαϊκές σχέσεις και κάπου, ε, χώρες, συγγνώμη, και κάπου θα πρέπει να αναφέρεται αυτό. Επίσης, θα έγραφα και κάτι άλλο. Ε, υπάρχουν στρατηγικοί και εταίροι μας που είναι η Βραζιλία και το Μεξικό. Εκτός από τον μπλοκ αυτό όλων των χωρών, ξεχωρίζουν οι δύο χώρες, Μεξικό και Βραζιλία και θα έδινα και μεγαλύτερη φιλοδοξία ε, σε αυτό που λέει ο Σαλαφράγκα για το Μεξικό. Λέτε να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις. Εξ όσων γνωρίζω έχουν αρχίσει. Αυτό που θέλουμε είναι να ολοκληρωθούν φέτος. Βέβαια έχουν παγώσει οι ε, διαπραγματεύσεις για το TTIP, ε, οπότε ανοίγει ο δρόμος για την Ιαπωνία, το Μεξικό και τη Χιλή. Μπορούν οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αφιερωθούν σε αυτές. Στο 18 δεν μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που λέτε, στο 5 χρειάζεται μια παράγραφος κάπου στην 5 να είναι πιο φιλόδοξη για τη σχέση μας. Η Σύνοδη Κορυφής με τη Λατινική Αμερική, στην παράγραφο 20 επειδή το παρακολουθώ αυτό το θέμα, έχουν ενισχυθεί αυτές, ε, Κάδι, ε, Βέρα Κρούς, Παναμάς, αναφέρω μόνο, και Γενική Γραμματεία, ε, όχι μόνο της Λατινικής Αμερικής, ολόκληρες της Νότιας Αμερικής, Ιμπεροαμέρικα, όχι η Λατινική Αμερική. Πρόεδρε, τελειώνω, τελειώνω. 22 δώστε μου. δεν χρειάζεται η, γραμματεία να εποπτεύει του έργου. Απλώς το πλαισιώνει, το συνοδεύει, το υποβοηθεί, αλλά δεν το εποπτεύει. Επίσης, ε, υπάρχει μια συμμαχία εκεί στον Ειρηνικό ε, που είναι παρατηρητές πολλές χώρες μέλη. Γιατί δεν ζητάμε από την κυρία Μογκερίνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Θα συνεχίσει να προεδρεύει ο κύριος Βίστησεν και νομίζω καλό θα ήταν να πει δύο λόγια ο εισηγητή για να κλείσει. Τρία-τέσσερα λεπτά, γιατί πρέπει να φύγω. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τα σχόλιά σας, για τις κριτικές και για τα όσα επισημαίνετε ε, για τις βελτιώσεις ή κάποιες ελλείψεις που μπορεί να έχει έκθεση για να προσθέσουμε ορισμένα πράγματα. Συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με τα όσα είπατε. Όλοι από όλες τις πολιτικές ομάδες. Να πω όμως μερικά πράγματα που μπορεί να βελτιωθούν κατά τις επόμενες εβδομάδες. Ακούσαμε από όλους μια ανησυχία για την κατάσταση στη Βενεζουέλα. Συμφωνώ. Το συζητήσαμε και τις τελευταίες εβδομάδες στο Κοινοβούλιο. Όταν εγώ εκπονούσα το κείμενο, τι είχα στο μυαλό μου ότι ταυτόχρονα έχουμε συζήτηση και ψήφισμα που εγκρίναμε την περασμένη εβδομάδα για τη Βενεζουέλα. Αυτή τη στιγμή εγκρίθηκε λοιπόν αυτό το ψήφισμα με ευρεία πλειοψηφία. Θα πρέπει να δούμε πώς εντάσσεται και πώς εγγράφεται στην έκθεση αυτό. Γιατί όντως είναι ανισχυτική η κατάσταση που επικρατεί εκεί. Αυτή ήταν ε, ε, η κεντρική μου ιδέα ότι υπήρχε μια παράλληλη διαδικασία για τη Βενεζουέλα και το Κοινοβούλιο και να περιμένουμε την έκβαση έλεγα και μετά να δούμε πώς θα το εντάξουμε στην έκθεση. Πολλά υπόθηκαν, πολύ εύστοχα. Εγώ θα ήθελα να επιμείνω σε μερικά. Ε, η διαφθορά, δικαιοσύνη, Ακούσαμε για την ελευθεροτυπία, πολύ σημαντικό και αυτό. Διάφοροι συνάδελφοι μίλησαν για το Μεξικό, για τη σημασία της Κούβας και τα εσωτερικά της προβλήματα, καθώς επίσης για τη γενικότερη κατάσταση στο Μεξικό που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τέλος, συμφωνώ ιδιαίτερα αυτά που είπε ο Ερνέστο Ουρτάσουν. Θα πρέπει να έχουμε κοινή πορεία στον ΟΗΕ και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς με τη Λατινική Αμερική. Είναι στρατηγικός εταίρος μας. Απολύτως. Αυτό μπορεί να είναι φιλοδοξία μας, γιατί δεν έχουμε μόνο κοινό όραμα, κοινή θεώρηση, αλλά έχουμε και κοινά θέματα, κοινή ατζέντα, που αυτό θα πρέπει να μεταφραστεί σε συνεργασία. Θεσμική, πολιτική, περιφερειακή, υπάρχουν τα εργαλεία. Και για το χρονοδιάγραμμα, ένα τελευταίο, τι είχαμε σκεφτεί για το φθινόπωρο, γιατί ακούσαμε από συναδέλφους ότι υπάρχουν διάφορα ζητήματα, διάφορα στοιχεία ε, που συμπίπτουν χρονικά. Εμείς θα θέλαμε να εγκριθεί η έκθεση πριν τη Σύνοδο Κορυφής. Και μετά τη Σύνοδο Κορυφής θα έρθει και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που έτσι είναι η λογική σειρά. Θέλω να σας θυμίσω κάτι που θα το γνωρίζετε. Μπορεί να υπάρχουν κάποια στοιχεία που να λείπουν από την έκθεση, σίγουρα θα έχουμε και λήψεις, αλλά ξέρετε ότι έχουμε περιορισμό χώρου στην έκθεσή μας και χαρακτήρων και δεν χωράνε όλα. Δεν μπορούμε να πούμε και τα περιφερειακά και ε, όλα όσα συμβαίνουν στη Λατινική Αμερική. Δεν θα χωράει αυτή η έκθεση. Αυτά. Ελπίζω και είμαι βέβαιος μάλλον ότι θα τη φέρουμε σε αίσιο πέρας. Ο κύριος Βίστησεν. Thank you to the Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε τον εισηγητή. Να σας ενημερώσω ότι η προθεσμία για την Κατάσταση τροπολογιών θα είναι στις 11 Μαΐου 12 η ώρα το μεσημέρι και έτσι ολοκληρώνουμε το σημείο αυτό στην ημερήσια διάταξη και περνάμε στα, στο 20, στα διάφορα. Δεν βλέπω τίποτε. Να σα ενημερώσω ότι η επόμενη συνεδρίαση θα λάβει χώρα 29 με 30 Μαΐου και έτσι ολοκληρώθηκε λοιπόν η σημερινή συνεδρίαση. Να περάσουμε τώρα στο εργαστήρι για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στην Μέση Ανατολή και στην ε, Βόρειο Αφρική και να προετοιμάσουμε παρακαλώ και την ένταση για